Good afternoon. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Ε, σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε θα ξεκινήσει τώρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους μου και τους διερμηνείς που είναι πολύ πληθέστεροι. και να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της κυρίας Σαρτόρη που μου ζήτησε να την αντικαταστήσω για την αρχή της συνεδρίασης. Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Και τώρα, αντί για Ιταλικά, έχετε Τσέχικα για αυτόν τον λόγο. Είναι μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις, συνεδριάσεις της ε, Επιτροπής μας αλλά είναι και μια έκτακτη συνεδρίαση. Πρώτο σημείο, η έγκριση της ημέρησιας διάταξης. Έχετε όλη την ημέρησια διάταξη. Εάν δεν υπάρξει κάποιο σχόλιο ή κάποια παρατήρηση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Ανακοινώσεις. Είναι κάπως τεχνικές οι ανακοινώσεις μου. Πρώτα απ' όλα. Έχει αλλάξει λιγάκι η για διάταξη, γιατί αύριο η συνεδρίαση από η Ματινή δυστυχώς έχει ακυρωθεί. Οπότε αύριο 18 θα έχουμε μόνο το πρωί συνεδρίαση. Δεύτερον, όπως ίσως ξέρετε, υπάρχουν νέοι κανόνες σε σχέση με την τελική ψηφοφορία στις Επιτροπές. Αυτό ετέθη σε εφαρμογή από τις 10 Φεβρουαρίου και φυσικά θα ισχύει και στην σημερινή συνεδρίαση και την αυριανή. Οπότε οι ψηφοφορίες αύριο γίνονται επί τη βάση των νέων κανόνων. Όλες οι τελικές ψηφοφορίες για τα ψηφίσματα θα γίνονται με ονομαστική κλίση. Οπομένω θα είναι <clears throat> ονομαστικές και ηλεκτρονικές. Πρέπει να έχετε την κάρτα σας μαζί σας. Όλες οι τελικές λοιπόν αύριο είναι ηλεκτρονικές και ονομαστικές. Κάτι ακόμα. Όταν τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση, παρακαλώ πάρτε όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα, γιατί ακολουθεί μια άλλη συνεδρίαση στις 7 ε, της ομάδος ε, των φιλελευθέρων. Οπότε μην αφήσετε τίποτα εδώ πέρα. Τέλος, τελευταία παρατήρηση. Αύριο στις 10 η ώρα, πριν από την ψηφοφορία δηλαδή, θα φωτογραφθεί η Επιτροπή μας ώστε να έχουμε αυτό το ιστορικό έγγραφο το οποίο θα αποδείξει ότι κάποτε εργαστήκαμε εδώ. Μία ομαδική φωτογραφία. και εφόσον ενδιαφέρεστε μπορεί να υπάρξει και ατομική φωτογράφηση από ό,τι πληροφορήθηκα. Αλλά μου είπε ο κύριος Κουάδρας ότι πρέπει να είσαστε καλά προετοιμασμένοι για τη φωτογραφία. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που έχετε φυσικά για τις κυρίες, αλλά όχι για τους άντρες. Λοιπόν, να έρθετε χαμογελαστία Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Έχουμε τα πρακτικά της 22ης-23ης Ιανουαρίου, καθώς και αυτά της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου. Έχουν διανεμηθεί τα έγγραφα αυτά μαζί με τα άλλα έγγραφα εργασίας. Εκτός εάν υπάρξει κάποιο σχόλιο ή κάποια αντίρρηση, θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί. και θα δημοσιευθούν ως έχουν. Αυτές είναι λοιπόν οι τεχνικές ανακοινώσεις που ήθελα να σας κάνω και ερχόμαστε τώρα στο τέταρτο σημείο που είναι το πρώτο ουσιαστικό σημείο στην ημερησία διάταξη. Είναι οι τροπολογίες στην οδηγία για την ποινική ασφάλεια ...215 τροπολογίες έχουμε μέχρι στιγμής έχουμε συμβαστικές τροπολογίες 7 τον αριθμό. Προβλέπετε μία ώρα για τη συζήτηση του θέματος αυτού και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Ρωμάνα Γιόρνταν ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε την άποψή της για τις τροπολογίες. Βέβαια ήταν πολλές τροπολογίες και της δίνω το λόγο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει λάβει η χώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, πήραμε 215 τροπολογίες. Καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων. Θα ήθελα πάντως να πω εξ αρχής ότι είχαμε μια καλή ε, ατμόσφαιρα εργασίας μεταξύ μας οι και γι' αυτό έχουμε προετοιμάσει 7 συμβιβαστικές. Ελπίζω ότι όλοι θα καλυφθούν εν μέρη. Βέβαια κάποια πράγματα δεν έχουν περάσει, αλλά αυτή είναι ακριβώς και η φιλοσοφία των συμβιβαστικών τροπολογιών. Πάντως γενικά νομίζω ότι έχουμε βρει κάποιο τρόπο έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ισχύουσα οδηγία. Στην πρώτη συμβιβαστική, την Α, είναι κάτι το οποίο λέει ότι το reasonably achievable, το έλογα εφικτό, έχει γίνει πρακτικά εφαρμόσιμο. Νομίζω ότι τη σωστή διατύπωση θα τη δείτε γραμμένη. Η δεύτερη συμβιβαστική αφορά την διαφάνεια έγκαιρη προειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση, άμεση ενημέρωση του κοινού. Η συμβιβαστική αυτή περιλαμβάνει επίσης η ενημέρωση του κοινού να καλύπτει όλα τα πεδία που έχουν σημασία από την έβρεση του χώρου μέχρι την θέση σε λειτουργία και φυσικά οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι συνέπειες της σύμβασης του Άρχου που επικαιρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι από την Ερατόμα, αλλά ξέρουμε ότι έχει σημασία η σύμβαση του Άρχου. Οι συμβιβαστικές 3 και 4 είναι οι στόχοι στον τομέα της ασφάλειας και εδώ έχουμε καταλήξει σε μια πιο συγκεκριμένη διατύπωση. Είναι περισσότερο κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες βέβαια εδώ. Η συμβιβαστική 5 αφορά την περιοδικό έλεγχο ασφαλείας. Αυτός ο περιοδικός έλεγχος είχε ήδη ζητηθεί και από την ισχύουσα οδηγία προσθέσαμε εδώ ότι τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουν οι αρχές προστασίας θα πρέπει να εφαρμόζονται πριν δοθεί άδεια για παράταση λειτουργίας. Η συμβιβαστική 6 τώρα για τα κατεπήγοντα προγράμματα αντίδρασης. Εδώ λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αναθεώρηση των προγραμμάτων ανά 8 ετία. Και στο τέλος είναι η συμβιβαστική για τον έλεγχο από ομολόγους. Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου από ομολόγους, όργανα και πρόσωπα το πρώτο αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και τα NRA και το δεύτερο αφορά τις τοπικές ε, τέτοιες αξιολογήσεις. Εδώ δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία και γι' αυτό υπάρχουν δύο συμβιβαστικές, η 7α και η 7β. Η 7α την προσυπογράφων η Φιλελεύθερη, το ΕΛΚ και η Πράσινη και την 7Β, ε, η EFD και η συντηρητική. Και στις δύο αυτές τροπολογίες το κείμενο είναι σχεδόν το ίδιο. Αλλά έχει σημασία στο ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι ε, βαρύτερος, ισχυρότερος. και είπαμε ότι θα πρέπει να καθοριστεί και στα πλαίσια της ΕΝΣΛΕΚ, της ομάδας δηλαδή των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας. Στην 7α υπάρχει ένας πιο σημαντικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα για τα θέματα της εξαετίας, και λέγει η Συμβιβαστική 7 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη γι' αυτό, ενώ η 7β δεν προβλέπει κάποιον τέτοιο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω επίσης ότι θα προτείνω τρεις προφορικές και στα πλαίσια των συμβιβαστικών αναθεωρήσαμε εμείς την αιτιολογική μας έκθεση και νομίζω ότι μπορέσαμε καθορίσουμε πιο σωστά τον ρόλο της ΕΝΣΕΛΕΚ. Θα συμπεριληφθεί λοιπόν στις αιτιολογικές σκέψεις. Συζητήσαμε και το θέμα της αλλαγής της νομικής βάσης Ζήτησα και γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και θα μας δώσει τη γνωμοδότησή της στις 20 Μαρτίου, όχι πριν την ψήφο, δηλαδή τη δική μας. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους συνεπώς να σεβαστούμε το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει σήμερα. Μπορεί και να διαφωνούμε με αυτό ίσως κάπου, αλλά σύμφωνα όμως και με την ιδρυτική συνθήκη, είναι σαφές ότι η νοβική ε, βάση εντάσσεται στη συνθήκη Αρατόμ. Θα συμφωνήσω βέβαια μαζί σας ότι θα πρέπει να δώσουμε μάχη για να αυξήσουμε το ρόλο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να βελτιώσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Και μια τελική παρατήρηση. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι άλλαξε η ημερομηνία της ψηφοφορίας από τον Απρίλιο 2 στον Απρίλιο 1, στην πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου. Ελπίζω να ψηφίσουμε λοιπόν στην πρώτη Ολομέλεια του μηνός Απριλίου. Ευχαριστώ λοιπόν την γραμματεία, ευχαριστώ τους συναδέλφους. για τη βοήθειά τους, την αίσθηση συνεργασίας τους και περιμένω τα σχόλιά τους πιθανώς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζόρνταν. Τώρα, θα περάσουμε στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις συζητητές, γιατί συμμετείχαν στις περίπλοκες συζητήσεις που έγιναν για να καταλήξουμε στις τροπολογίες αυτές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο κύριος Κορέτ Κάμπος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, πράγματι, πολύ χαίρομαι που εσείς προεδρεύετε εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω και σας αλλά και την κυρία Τζόρνταν, την κυρία Ρωμάνα Τζόρνταν για την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε και έτσι μπορέσαμε να συζητήσουμε στις διάφορες συναντήσεις πολύ καλά μεταξύ μας. Την ευχαριστώ επίσης και για την σταθμισμένη της στάση σε σχέση με την νομοθετική αυτή πρόταση. Η αναθεώρηση της οδηγίας αυτής είναι κάτι αναγκαίο και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία που παίρνουμε μετά το ατύχημα στο Φουκουσίμα. Τα μαθήματα που πήραμε μετά από το φοβερό αυτό ατύχημα και όλα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν σε νέους νόμους, σε νέες πρακτικές για να αυξηθεί η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Αυτό που προτείνει η οδηγία δεν είναι τόσο ιδιαίτερα φιλόδοξο όσο θα μπορούσε να είναι. Ούτως ή άλλως όμως αναγνωρίζουμε ότι η πρόταση αυτή είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για τα θέματα της ποινική ασφάλειας και φυσικά δεν είναι εύκολο να επιτύχει κανείς ριζική πρόοδο. Ο τομέας ποινική ενέργειας είναι και ένας χώρος όπου τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών πολλές φορές έχουν μια συντηρητική χρειά και προτιμούν να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη αυστηρότητα στους κανόνες ασφάλειας και επομένως υπάρχει μια αντιπαράθεση απόψεων η οποία αντανακλάται και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από αυτή την πλευρά οι διαπραγματεύσεις που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα οδήγησαν σε μια συμφωνία για 8 τροπολογίες συμβιβασμού. Κατά την απόψή μας είναι ισορροπημένες αυτές οι τροπολογίες και η σοσιαλιστική ομάδα προσπάθησε μέσα από αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες να διατηρήσει και να ενισχύσει πάντα την πτυχή της ασφάλειας μέσα στην πρόταση της Κομισιόν και προσπάθησε να εξασφαλίσει και μεγαλύτερη ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστών για τον τομέα της ενέργειας. Η διαδικασία του peer review, της, ε, του ελέγχου από τους ομοτήμους, είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για να μπορέσουμε να βγούμε από τη σημερινή σύγχυση που επικρατεί με αντιμαχόμενα συμφέροντα των κρατών μελών και να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και ο αυξανόμενος ρόλος της Κομισιόν σε συντονιστικό επίπεδο, ο συντονιστή δηλαδή τους ε, των εθνικών ρυθμιστών και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος ότι πρέπει να γίνει πράγματι αυτός ο συντονισμός από την Κομισιόν. Υποστηρίζουμε επίσης και την τροποποίηση της νομικής βάσης του κανονισμού ε, από τη συνδίκη της Ευρατόμου στα αρμόδια άρθρα της συνδίκης της Λισαβόνας, διότι αυτό θα δώσει ρόλο ε, συναπόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα μπορεί έτσι να εξασφαλίσει περισσότερο τα θέματα ασφάλεια και υγείας σε ό,τι αφορά τα θέματα πυρηνική ενέργεια. Ε, Παρ' όλα αυτά, όπως ε, είπε και η συγγητρία, δεχόμαστε ότι εάν δεν υπάρξει άλλη δυνατότητα, μπορεί η συζήτηση να γίνει μέσα στα πλαίσια της ε, Ευρατόμ. Κλείνοντα, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τι προσπάθειε τη, που ήταν πάρα πολύ σημαντικέ και πάρα πολύ χρήσιμε, και θέλω να πω ότι από την πλευρά των σοσιαλιστών και δημοκρατών δεν βλέπουμε κανένα ρόλο να μην δώσουμε θετική ψήφο στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τεκάμπος, ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε. Δεν έχουμε εδώ όλους τους σκιώδεις, οπότε επιτρέψτε μου να μιλήσω κι εγώ. Κι εγώ θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέρφους τα συγχαρητήρια που έδωσαν στην εισηγητριά μας είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα. Υπήρξαν πολλές διαφορετικές απόψεις, αντίθετες μεταξύ τους μερικές φορές. Οι χώρες μέλη από την άλλη μεριά έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τα, τους πυρηνικούς σταθμούς και την ασφαλειά τους. Συνεπώς δεν ήταν καθόλου εύκολο να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Συνεπώς, είναι κατανοητό μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα να γίνονται πολύ έντονες συζητήσεις όσον αφορά την ασφάλεια από τα πυρηνικά και δεν είναι εύκολο βέβαια κανείς να αποφανθεί σε σχέση με την προτινόμενη οδηγία. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Τζόρνταν, η οποία ε, πράγματι προσπάθησε να καταλήξει σε λύση, παρόλο που οι απόψεις ήταν συχνά πολύ διαφορετικές μεταξύ μας. Είναι μεγάλο επίτευγμα δηλαδή που τα κατάφερε να φτάσει σε τροπολογίες συμβιβασμού. Εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας μπορώ να πω ότι είναι ζωτική σημασίας να στηρίξουμε και να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής. Οι εθνικοί επιθεωρητές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και πραγματικά επαγγελματίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών είναι ζωτική σημασία για μας. Συνεπώ, όσον αφορά τι έξι πρώτες τροπολογίες, συμφωνώ με την εισηγήτρια και δεν βλέπω εδώ να υπάρχει τίποτα το επίμαχο ή κανένα πρόβλημα. Εκεί που διαφέρει η δικιά μας η άποψη είναι στο θέμα της, ε, του ελέγχου από τους ομόλογους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει το ρόλο διαιτητή κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε να το διατυπώσω έτσι. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Η δικιά τους η άποψη είναι ζωτική σημασίας και οι δικές τους οι απόψεις πρέπει να εισακούονται και να χρησιμοποιούνται. Το πιο σημαντικό λοιπόν για μας είναι η επικοινωνία μέσα στην ΕΣΡΕΚ και όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία εκεί θα δείτε τη δικιά μας την άποψη. Γι' αυτό υπάρχει 7α και 7β και οι δύο τροπολογίες θα υποβληθούν χωριστά για ψηφοφορία αύριο. Αυτό είναι ένα θέμα σχετικά με το οποίο δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να υποβάλουμε δύο διαφορετικές τροπολογίες, δύο ξεχωριστές τροπολογίες πιο σωστά. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι την εισηγητριά μας, την κυρία Τζόρνταν. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και για την ικανότητά σας να καταφέρετε να συμβιβάσετε τις απόψεις μας. Ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λογική λύση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η δικιά μου άποψη. Δεν βλέπω κανέναν άλλο σκιώδη συγκητή εδώ. Συνεπώς μπορούμε να συνεχίσουμε και να αρχίσει η συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Γκροστέτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, εδώ πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύ ευαίσθητο. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγητριά μας. Η δουλειά που έκανε ήταν ε, περίπλοκη, δύσκολη για να καταφέρει να συγκεντρώσει και να συμβιβάσει θέσεις που συχνά απόκλειναν μεταξύ τους και μάλιστα για ένα θέμα ζωτικής σημασίας όπως είναι η αναθεώρηση αυτή. Όσον αφορά την νομική βάση πρώτα απ' όλα, είναι ένα θέμα που επανέρχεται και το γνωρίζω από τότε που πρωτοήρθα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επανέρχεται σε όλες τις εκθέσεις που έχουν να κάνουν με την πυρηνική ενέργεια. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να διατηρήσουμε την νομική βάση γύρω Euratom. Είναι πολύ επικίνδυνο να ξανανοίξει η συζήτηση αυτή, διότι τότε θα καταλήγαμε σε μια πολύ βαριά διαδικασία, θα χρειαζόταν μια διακυβερνητική διάσκεψη, ομοφωνία και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να υπάρξει τέτοια προσέγγιση στα πλαίσια της αναθεώρησης αυτές της οδηγίας. Δεύτερον, για τη διαφάνεια. Φυσικά και όλοι συμφωνούμε Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και συμφωνώ με τις προτάσεις που έχουν στόχο να βελτιώσουν τη διαφάνεια αυτή απέναντι στους πολίτες μας για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες τους, στις απορίες τους. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην πυρηνική ενέργεια που είναι ζωτική σημασία για την ενεργειακή αυτονομία και προκειμένου να χρησιμοποιούμε λιγότερο άνθρακα στην οικονομία μας. Μέχρι τώρα τα πυρηνικά υπέφεραν από μια πολύ κακή εικόνα που είχαν εξαιτία τη κακή επικοινωνία και εξαιτία του ότι δεν υπήρχε διαφάνεια. Δεν ξέραν οι πολίτε. Οπότε πρέπει να υπάρξει πρόοδο στον τομέα τη διαφάνεια. Τρίτον, κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Και εδώ συμφωνώ μαζί σας, Πρόεδρε. Γιατί ένα από τα μαθήματα που πήραμε με το ατύχημα της Φουκουσίμα είναι ότι ο ρυθμιστής δεν είχε στη διάθεσή του αρκετή εξουσία πάνω σε αυτόν που εκμεταλλεύεται τον πυρηνικό σταθμό σε σχέση με την ασφάλεια και δεν μπορούσε να έχει αποτελεσματικό έλεγχο. Και γι' αυτό και στηρίζω τις τροπολογίες που θέλουν να ενισχύσουν την ανεξαρτησία, την αυτονομία των αρχών αυτών των εθνικών για την ασφάλεια. Είναι απαραίτητο οι αρχές αυτές να έχουν και τα νομικά και τα οικονομικά μέσα για να είναι ανεξάρτητες αρχές σε σχέση με τις υπόλοιπες εθνικές αρχές και τα διάφορα λόμπις. Γι' αυτό όμως ανησυχώ για κάποιες τροπολογίες όπως και για τη συμβαστική τροπολογία 7α. Αποδυναμώνει για να μην πω ότι βγάζει παντελώς την ευθύνη από τους ώμους των ε, εθνικών αρχών και την μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε ήδη εγκρίνει ψήφισμα για την αξιολόγηση κινδύνων και για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών. Καταλήξαμε σε έναν απολογισμό μετά από δοκιμές που έγιναν αντοχής και που τις έκανε η Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εναρμόνιση στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεβάζοντας τις προδιαγραφές, τονίζοντας ακόμα περισσότερο τις ανταλλαγές που πρέπει να υπάρχουν όσον αφορά την ενημέρωση και την αύξηση των μηχανισμών ελέγχων. Γι' αυτό όμως πρέπει η ΕΝΣΡΕΚ να παρεμβαίνει περισσότερο να εμπλέκεται περισσότερο και να χρησιμοποιεί και επιπλέον επιστημονική πραγματογνωμοσύνη, όπως προτείνει η τροπολογία. Που την προτιμώ από την 7α, η οποία προτιμά να δώσει περισσότερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προτιμώ την τροπολογία 7β, που δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στις ρυθμιστικές αρχές. Συνεπώς, είπα για την ανεξαρτησία, μην επανέλθω σε αυτό. Είπα για τις αρχές της εθνικής ασφάλειας που πρέπει να είναι στην καρδιά της διάταξης, των διατάξεων που περιλαμβάνονται εδώ για την ασφάλεια. Οπότε κάθε ε, τροπολογία που αναφέρεται στον έλεγχο ομολόγων μέσω της ΕΝΡΕΝΚ με βρίσκει σύμφωνη. Πρέπει τα θέματα πυρηνικής ασφάλειας να είναι φιλόδοξη, παρακολούθηση να είναι αποτελεσματική και συγχρόνως όμως διατήρηση της ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας. Αυτά είχα να προσθέσω εγώ σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχεις δει στο λόγο ο κ. Βιντάλ Κουάντρας. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια προς την εισηγητρία η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ καλή δουλειά και επιπλέον αυτή τη στιγμή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία το έργο της γιατί χρειάστηκε να εργαστεί με μεγάλη ταχύτητα επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας και είναι στενές οι προθεσμίες και είναι απαραίτητο για να μην πάει στράφη το έργο μας στους τελευταίους μήνες πρέπει να κινηθούμε ταχαίω ώστε να προλάβουμε την τελευταία ολομέλεια. Συζητούμε τώρα τις τροπολογίες για να ψηφίσουμε αύριο. Όλα αυτά είναι απαραίτητα αν θέλουμε πράγματι να κλείσουμε όλα αυτά τα εκκρεμή θέματα τα οποία δεν θέλουμε να τα αφήσουμε για το επόμενο κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την υποστήριξή μου στις ε, τροπολογίες οι οποίες αναγνωρίζουν το ρόλο, το σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές γιατί αυτοί είναι που έχουν τον, γνωρίζουν τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα τους, η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε να βελτιώνουμε την ασφάλεια στον τομέα αυτό που είναι τόσο κέριος. και πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να έχουν ανεξαρτησία οι ρυθμιστές, οι εθνικοί ρυθμιστές και φυσικά να έχουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας. Γι' αυτό το κάθε κράτο θα πρέπει να είναι προσεκτικό στον τρόπο με τον οποίο ε, διορίζει αυτά τα άτομα. Δεν πρέπει να γίνονται πολιτικοί διορισμοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τα τεχνικά και επιστημονικά ε, κριτήρια. Αυτό είναι κρίμα λοιπόν να γίνεται, γιατί πρέπει οι ρυθμιστές να είναι άτομα υψηλών προσόντων από αυτούς οι οποίοι έχουν ε, καθήκοντα καθημερινού ελέγχου μέχρι αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας, όλοι τους θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές γνώσεις για τον τομέα αυτό. Αυτό λοιπόν ιδιαίτερα θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε και γι' αυτό καταθέσαμε και μια τροπολογία γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη όπου δυστυχώ οι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια ελαφρά την καρδία διορίζουν τον πρώτο που βρίσκουν με κριτήρια καθαρά πολιτικο-κομματικά. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο κρίμα. Ένα πρόβλημα της ε, πυρηνικής βιομηχανίας είναι πάντα η στάση της κοινή γνώμης. Εδώ είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομπρέλα για την πυρηνική ασφάλεια δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο κοινό και έτσι ευνοεί την εξέλιξη του τομέα αυτού και θέτει ένα ανάχωμα στους λαϊκιστές και στους δημαγωγούς. Τούτου λεχθέντος είναι αλήθεια ακόμα ότι η Ευρατόμ είναι η συνθήκη που διέπει τα πυρηνικά, αλλά το μείγμα ενέργειας είναι θέμα εθνικής απόφασης και φυσικά η πυρηνική ενέργεια έχει στρατηγική έχει στρατηγικό χαρακτήρα για τις χώρες που την χρησιμοποιούν. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει απόλυτο σεβασμός αυτών των εθνικών επιλογών. Νομίζω λοιπόν ότι όλα είναι έτοιμα για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή ψηφοφορία αύριο και η κυρία Γιόρταν μπορεί να νιώσει ανακούφιση και να ξέρει ότι οι προσπάθειές της έχουν οδηγήσει σε μια πολύ ψηλή ποιότητα εργασίας όπως και περιμέναμε από αυτήν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Η κυρία Χιούμπνερ θέλει να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές ότι το ατύχημα της Φουκουσίμα μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλεια είναι αυτή η οποία θα πρέπει να έχει τον καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη στα πλαίσια της συζήτησης για τα πυρηνικά και εξ αυτού προήλθε και η εξαιρετική ε, πρόταση της συναδέλφων. Στην έκθεση αυτή υπάρχει αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Θελήσαμε πράγματι να υπάρξει μια σωστή παρακολούθηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων, να υπάρξει ένα σαφής έλεγχος όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αναφερθήκαμε επίσης και στην ανάγκη ύπαρξης ενός πλήρους ελέγχου στα πλαίσια των κύκλων περιοδικού ελέγχου. Αυτό θα επιτρέψει να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Τρίτον, αναφερθήκαμε στο ότι τα ελεγκτικά όργανα όλων των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτυχθούν σωστά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, πιθανότητες, να μειωθούν οι πιθανότητες ατυχημάτων. Τώρα, σε επίπεδο πρακτικό. Πού βρίσκεται η κατάσταση σήμερα στις συζητήσεις. Ε, θα μπορούσαμε να υπονομεύσουμε τις αρχές ε, ή μάλλον τις δυνατότητες, τις αρμοδιότητες των οργάνων αυτών. Αυτό δεν θα ήταν σωστό γιατί καλά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν πρέπει να θέσουμε σε αμφισβήτηση την ύπαρξή τους και τη λειτουργία τους. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τη δράση τους και δεν θα πρέπει να ακούγονται κριτικές σχετικά με τις αρμοδιότητες τους και τις ικανότητες τους. Αυτό που είπε η Φρανσουάζ έχει σημασία. Στο μέλλον είναι βέβαια σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε εναρμονισμένα κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα καθορίσουμε κάποια ανώτατα όρια γύρω από τα θέματα της πυρηνικής ασφάλειας. Αυτός είναι ο στόχος μας λοιπόν για το μέλλον και ελπίζω να τα συζητήσουμε αυτά εκ νέου και να προετοιμάσουμε τη σωστή νομοθετική ρύθμιση που θα μας διευκολύνει. Πάντως έχει φτάσει πλέον η στιγμή να προωθήσουμε το διαφορετικό ενεργειακό μίξ αναχώρα, λαμβάνοντας υπόψη και τον πυρηνικό τομέα δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι η πυρηνική ενέργεια είναι κακή και απαράδεκτη κοινωνικά. Δεν ισχύει αυτό. Να εξηγήσουμε τα προβλήματα ασφαλείας τα οποία μπορεί να υπάρχουν και να τους εξηγήσουμε ότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος είναι ασφαλής και για την υγεία των πολιτών και διασφαλίζει φτηνή και καλή ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα συμφωνήσω με αυτούς που ευχαρίστησαν την κυρία Ιορντάν για την ε, δουλειά την οποία έχει κάνει. Είναι περίπλοκο το θέμα. Για τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας δεν έχουμε διαιρέσεις μεταξύ μας σε πολιτικό επίπεδο εκτός ίσως από τους πράσινους, αλλά ε, βασικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε χώρες. Χώρες είναι υπέρ της παραγωγής, άλλες χώρες είναι κατά. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω τα μέτρα τα οποία οδηγούν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών Υποστηρίζω επίσης την αύξηση των επιπέδων διαφάνειας με στόχο αυτό το οποίο θα ονόμαζα καθ' η απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια. <coughs> Όμως Γνωρίζουμε ότι τίθεται εδώ το θέμα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επηρεάζει τις ρυθμιστικές αρχές και θα υποστηρίξω την τροπολογία 7β. Είναι εξαιρετική η δουλειά της συναδέλφου. Η συμβιβαστική αυτή πρόταση είναι μια εξαιρετική πρόταση γιατί όπως είπα από τη μία υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μου αρέσουν αλλά από την άλλη βλέπω ότι και οι αντίθελοι, οι αντίθετοι πιστεύουν ότι η συμβιβαστική πρόταση περιλαμβάνει θετικά στοιχεία και γι' αυτό θα την υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάσκα τώρα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Τζόρνταν για τη δουλειά της. Κατάφερε με πολύ υπεύθυνο τρόπο να φέρει σε πέρα στη δουλειά αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την νομική βάση της Euratom και πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να προχωρήσουμε με το νομοθετικό μας έργο. Επίσης πιστεύω ότι η θέση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ανεξάρτητη. Όσο λειτουργούν καλά οι διεθνείς κανόνες και έχουν αρμοδιότητες οι ρυθμιστικές εθνικές αρχές, τότε νομίζω ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι αναγκαία σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει δηλαδή να βασιστούμε στους διεθνείς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου, αλλά παντού. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος των ομιλητών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκαρίμπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι μετά από αυτά που ακούσαμε σήμερα, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από όλες τις πτέρυγες για το θέμα αυτό και αυτό ικανοποιεί ιδιαίτερα την Κομισιόν. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω το έργο του εισηγητή γιατί στάθηκε ικανός η συγγήτρια, γιατί στάθηκε ικανή να συγκεράσει τις διάφορες απόψεις και να μειώσει τις ε, τροπολογίες, τον αριθμό των τροπολογιών σε 7 ή 8 συμβαστικές τροπολογίες, ξέρετε πώς βλέπετε τον κατάλογο. Θα επίσης να υπογραμμίσω ότι, να πω επίσης ότι η χρονική στιγμή της απόφασης που θα πάρετε είναι μεγάλη σημασία γιατί όπως υπογράμμισαν κάποιοι ομιλητέ, το νομοθέτημα αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της απάντησης που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα γεγονότα της Φουκουσίμα. Γι' αυτό είναι ζωτικό το τρέχον κοινοβουλίο και όχι το επόμενο να εκφέρει γνώμη σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν ώστε να μπορέσει να κλείσει ο φάκελος των θεμάτων αυτών το ταχύτερο δυνατό. Και φυσικά αυτό είναι ένα επίτευγμα το ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο και στη... τον έπαιρνο γι' αυτό πρέπει να πάρει η συγγήτρια αλλά και όλες οι συγγητές οι οποίοι έδειξαν μια ιδιαίτερα επικοδομητική στάση για το θέμα αυτό. Επίσης να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες εμείς έχουμε κάνει μια αρκή, αρχική έχουν δώσει μια αρχική ματιά σε όλες τις τροπολογίες και μπορώ να σας πω ότι η Κομισιόν υποστηρίζει πλήρως ή εν μέρη όλες τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατέθει και δεν θα σας εκπλήξει ότι μεταξύ της 7α και της 7β η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμάει λίγο περισσότερο την 7α. Η, η άλλη συζήτηση η οποία έχει αναφερθεί κατ' επανάληψη στην ε, Επιτροπή σας είναι το θέμα της νομικής βάσης για αυτή την πρόταση. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι κατανοούμε μεν τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις νομικές βάσεις για την συνθήκη της Ευρατόμ αλλά στο συγκεκριμένο αυτό νομοθέτημα πρέπει να σας υπενθυμίσω δύο γεγονότα. Πρώτα ότι το 2002 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενέκρινε ως ε, νομική βάση για τα ποινικά θέματα το άρθρο 31 και επέκεινα της ε, Συνδίκης Ευρατών και δεύτερον εφόσον εδώ έχουμε μια τροποποίηση προηγούμενης οδηγίας που ήδη βασίζεται σε συγκεκριμένα άρθρα της συνθήκης ε, Ευρατόμ από την πλευρά της Κομισιόν είναι προφανής η επιλογή της συνεκτικότητας και επομένως της διατήρησης της νομικής βάσης. Του τουλεχθέντος βέβαια, νομίζω ότι η συγγήτρια έχει παρουσιάσει ήδη την ανάλυση των τροπολογιών. Ναι, τονίσω εγώ από τη δική μας πλευρά ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η κύρια ιδέα που διατρέχει την τροποποίηση της οδηγίας, δηλαδή η ανεξαρτησία των ρυθμιστών, η μεγαλύτερη διαφάνεια, το μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, όλα αυτά γίνονται απόλυτα δεκτά από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ λέγει ο Πρόεδρος. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στην εισηγέτρια για να συνοψίσει τη συζήτηση. Έχετε το λόγο κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ. Υπάρχει διερμηνία στα σλοβενικά, οπότε θα συνεχίσω στα σλοβενικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Όλους παρακολούθησα τη συζήτηση και θα ξεκινήσω με τη νομική βάση, το θέμα της νομικής βάσης. Πράγματι θα ήθελα να ελπίζω η νομική βάση να μην μας δημιουργήσει προβλήματα και να μην αφήσουμε το θέμα για εξέταση από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το ατύχημα της Φοκουσίμα συνέβη στην αρχή της εντολής μας και οφείλουμε στους πολίτες μας να αντιδράσουμε τώρα. Το να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση για την νομική βάση αυτό σημαίνει κολυσιεργία. Το θέμα δεν είναι ότι δεν είναι σαφές ότι εμείς υιοθετούμε μια νέα οδηγία, αλλά στην ουσία τροποποιούμε την οδηγία η οποία έχει διατυπωθεί αρχικά βασισμένη στην συνθήκη ερατών. Χαίρομαι που είμαστε ομόφωνοι σχετικά με τα θέματα ασφαλείας. Χαίρομαι επίσης ότι όλοι ε, βάζουμε σαν πρώτο βασικό ε, θέμα το θέμα της ασφάλειας. Πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε ακριβώς αυτό και να ε, ε, προβλέψουμε τους απαιτούμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να λειτουργήσουν σωστά οι μηχανισμοί ασφαλείας. Αναφερθήκατε επίσης στην ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Άποψή μου είναι ότι η 7α επιτρέπει να υπάρξει με σωστό τρόπο η ανεξαρτησία αυτή. Σύμφωνα με τη νέα διατύπωση, οι νέες ρυθμιστικές αρχές θα έχουν την ανεξαρτησία την οποία επιθυμούν. Η διαφορά είναι μόνον η εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορισμένες αρμοδιότητες σχετικά με αυτό και αυτή είναι μια διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και συνεχίζει να ισχύει και στην περίπτωση των τεστ αντοχής, των δοκιμών αντοχής. <clears throat> Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να απομονώσουμε τις εκτιμήσεις για την ασφάλεια στα κάθε κράτος μέλος. Η ΕΝΣΟΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήκει σε αυτήν θα πρέπει να συναντάτε και να αποφασίζει για το πώς θα εφαρμοστούν οι συστάσεις αυτές. Δεν έχει σημασία εάν θα υπερψηφίσουμε το 7α ή το 7β, όπως και να έχουν τα πράγματα βελτιώνουμε την οδηγία, αλλά εγώ σαν εισηγήτρια εμένω στην 7α. Θα ήθελα λοιπόν για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία σας, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους άλλους και τη γραμματεία και τους ε, απλούς συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν απολύτως δεκτική απέναντί μας, οπότε θέσαμε ερωτήσεις, μας απάντησε έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση που προηγήθηκε. Τελειώνει μια μακρά συζήτηση θα έλεγα μεταξύ των σκιωδών και των εισηγητών. Σας ευχαριστώ όλους για τις προσπάθειές σας. Όπως είπε και ο Βιντάλ Κουάντρας δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή. Θυμίζω ότι θα ψηφίσουμε την έκθεση Γιόρνταν αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί μετά τις φωτογραφίσεις. Πρώτα θα μας φωτογραφίσουν και μετά θα ψηφίσουμε. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα, τη συζήτηση με τον κύριο Ντομινί Κριστόρη τον νέο Γενικό Διευθυντή της DG στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό λοιπόν τον κύριο Ριστόρη να έλθει εδώ. Ještě Καλώς ήρθατε και πάλι. Κύριε Ριστόρη, καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής μας. Είναι τιμή για μας να σα έχουμε εδώ μαζί μας για να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα μιλήσουμε για ένα τεράστιο εύρος θεμάτων σχετικών με την ενέργεια. Όλοι γνωρίζουμε στην Επιτροπή μας η ενέργεια είναι το κυρίως θέμα που συζητάμε και που θα συζητάμε στο μέλλον. Είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας και πολύ ενδιαφέρον για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως Είδαμε και στη συζήτηση που κάναμε μόλις πριν, δεν είναι εύκολο το θέμα, γιατί κάθε χώρα μέλος έχει μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα που θέλει να χρησιμοποιεί, γιατί αυτό εξαρτάται από το ιστορικό και το πολιτιστικό υπόβαθρο. Κύριε Γενική Διευθυντά, καταλαβαίνατε ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάντως που ήρθατε εδώ και παρακαλώ σας δίνω και το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ριστόρη. Κάντε μας μια εισαγωγή και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ και μάλιστα η στιγμή αυτή συμπίπτει με μία επικαιρότητα όπως το υπενθυμίσατε και εσείς που πάλι την ενέργεια την βάζει στο κέντρο της πολιτικής μας προσοχής και ενδιαφέροντος. Αυτό ισχύει για την Ευρώπη, αλλά όχι μόνο. Ισχύει και διεθνώς, γεωπολιτικά μιλώντας δηλαδή. Επιθυμώ λοιπόν, μέσα από την παρέμβασή μου αυτή, να υπογραμμίσω κυρίως δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα όσον αφορά το διεθνές, το παγκόσμιο πλαίσιο η Ευρώπη δεν είναι μόνη της στην ενέργεια, εννοείται ότι πρέπει να λάβει υπόψη της τις εξελίξεις, τις αλλαγές. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι από εκεί εννοείται ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας πρέπει να σχεδιαστεί βάσει μια σωστή ισορροπίας, right balance, ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα που θέλουμε και την βιωσιμότητα. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με αυτά που αλλάζουν στη διεθνή σκηνή και όχι μόνο για μας. Υπάρχει διαφοροποίηση πηγών πρώτα απ' όλα. Όλο και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Και από την άλλη μεριά, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μη συμβατικά, ιδίως στις Ηνωμένε Πολιτείες, με επιπτώσεις επί των τιμών και επί της ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον, βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη πίεση στη ζήτηση. Και κατά τη γνώμη μου είμαστε μόνο στην αρχή. Γιατί υπάρχει ένα τριπλό εδώ θέμα. Έχουμε την δημογραφική εξέλιξη. Βλέπουμε να επιταχύνεται ε, φοβερά η δημογραφική πρόοδος. Ένα δισεκατομμύριο θέμαστε σε λίγο και μετά βλέπουμε ότι το 2063 7 δις. Καταλαβαίνετε ότι η πρόοδος η δημογραφική είναι τεράστια. Δεύτερον, όσον αφορά με το τι ασχολείται ο πληθυσμός αυτός. Ήταν κυρίως αγροτικός ο πληθυσμός, τώρα κυρίως βρίσκεται στις πόλεις και η ενεργειακή όρεξη του πληθυσμού αυτού πολλαπλασιάζεται. Τρίτον, έχουμε πολύ γρήγορη εξέλιξη της ε, μεσαίας τάξης, που είναι όλο και πιο πολύ αριθμοί. Τις δύο επόμενες δεκαετίες, 2 με 3 δισεκατομμύρια παραπάνω άνθρωποι θα μπουν στην κατηγορία αυτή της μεσαίας τάξης, κυρίως στην Ασία, Κίνα, Ινδία, αλλά και στην Λατινική Αμερική και την Αφρική. Συνεπώς μπορούμε να προβλέψουμε επιπτώσεις επί των τιμών που θα είναι πολύ σημαντικές τιμές που θα παραμείνουν υψηλές για την ενέργεια. Και το τελευταίο στοιχείο, που δεν είναι ουδέτερο και αυτό και απορρέει από την ανάλυση αυτή, είναι ο ανταγωνισμός όλο και περισσότερο γεωπολιτικά ανάμεσα στις διάφορες οικονομικές δυνάμεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους. Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που και αυτή ενισχύει το όλο και περισσότερο για τις αγορές. Γιατί είχαμε μόνο το πετρέλαιο ως παγκόσμια αγορά, ενώ τώρα βλέπουμε να ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για το φυσικό αέριο και για το εγροπημένο φυσικό αέριο, αλλά και για το μη συμβατικό. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, εμείς που έχουμε τόσο λίγους πόρους, χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική, λαμβάνοντα υπόψη την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και βέβαια την ε, ενεργειακή ασφάλεια. Και εδώ υπάρχουν διάφοροι άξονε γύρω από του οποίου μπορούμε να στραφούμε. Ο πρώτο είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε τη χρήση του άνθρακα. Αλλά και αυτό ισορροπημένα, γιατί δεν υπάρχουν εδώ πέρα μόνο κακανέα. Πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα στην Ευρώπη έχουμε 50% του ηλεκτρισμού μας ήδη από σήμερα, 2014, έτσι δεν μιλάω για 2020 που παράγεται χωρίς διοξίδιο του άνθρακα. Με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σήμερα είμαστε στο 21-22% και την πυρηνική ενέργεια βέβαια. Ο συνδυασμός αυτός είναι 50% του ηλεκτρισμού χωρίς διοξίδιο του άνθρακα. Και είμαστε η πρώτη ζώνη στον κόσμο που το πετυχαίνει αυτό. Και ξέρετε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για το 2030 40% μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Και χαίρομαι εξάλλου που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε προς την ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Και διαπιστώνω ότι πολλές χώρες μέλη στηρίζουν το στόχο αυτό. Ακόμα βέβαια και αν παραμένουν κάποια ερωτηματικά με την Πολωνία και κάποιες άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είναι βέβαια θεμητά ζητήματα αυτά. Πρέπει συνεπώς να αναπτύξουμε περισσότερο τις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα γιατί ο άνθρακας θα συνεχίσει να υπάρχει και να χρησιμοποιείται για αρκετό χρόνο ακόμα στην Ευρώπη. 80% για την παραγωγή ηλεκτρισμού στην ε, Πολωνία. Αλλά θα χρησιμεύει και στις αναδυόμενες οικονομίες. Θα είναι κυρίαρχος ο άνθρακας. Άρα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να φροντίσουμε να έχουμε τέτοια τεχνολογία καθαρού άνθρακα σε επίπεδο Ευρώπης και επιχειρήσεων ευρωπαϊκών. Χρειαζόμαστε επίσης ανάπτυξη των αναλλακτικών πηγών ε, ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη μας την αγορά. Αυτό ακριβώς είναι που προτείνουμε με τον στόχο του 27% να συνοδεύεται όμως ο στόχος αυτός με τον στόχο της αγοράς, δηλαδή να συνοδεύεται από επιδοτήσεις οι οποίες να σταματούν όταν γίνεται εμπορικά βιώσιμη μια ενέργεια. Χρειαζόμαστε βέβαια ένα ισορροπημένο και διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα. Έχουμε λίγους ενεργειακούς πόρους στην Ευρώπη, οπότε εννοείται ότι δεν πρέπει να βάζουμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Πρέπει επίσης να υπάρξει η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς με ένα δίκτυο απόλυτα ενωπημένο. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό κάποιες χώρες μέλη να παραμένουν εξαρτώμενες από τρίτες χώρες. Οι βαλτικές χώρες, για παράδειγμα, που εξαρτώνται πλήρως από τη Ρωσία. Πρέπει επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στις διασυνδέσεις, τις ζώνες που χρειάζονται περισσότερο την βοήθεια. Στην Ιβυρική Χερσόνησο, για παράδειγμα, η σύνδεση Πυρηναία με τη Γαλλία είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε. Και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μίλησα με αρμόδιους από την Ισπανική και τη Γαλλική πλευρά. Χρειαζόμαστε επίσης μία ενισχυμένη περιφερειακή προσέγγιση. Και γιατί γιατί οι ίδιες συνδέσεις, η ανάπτυξη υποδομών δικτύων είναι κάτι το οποίο βέβαια προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο. Συνεπώς πρέπει πρώτα απ' όλα να χτίσουμε εκεί που ήδη υπάρχουν διασυνδέσεις, εκεί που υπάρχουν ενισχυμένες συνεργασίες ανάμεσα στις αρχές, τους ρυθμιστές, τα δίκτυα κλπ. Ιδιαίτερα εδώ αναφέρομαι στο βορρά και να λάβουμε υπόψη μας και το νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό τμήμα της Ευρώπης και να επικεντρώσουμε την δουλειά μας και τη δουλειά των ρυθμιστών στα κατά προτεραιότητα προγράμματά μας. Έτσι θα διαχειριστούμε καλύτερα την ε, συμπερίληψη των ε, νέων ενεργειών. Θα υπάρχει ένα τμήμα με κεντρική διαχείριση και ένα με αποκεντρωμένη και διαχειριστούμε έτσι καλύτερα τις ικανότητές μας. Περιφερειακά λοιπόν πρέπει να γίνουν αυτά. Τρίτον, πολιτική ζήτηση και κυρίως ενεργειακή απόδοση. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο από τα πιο προηγμένα να το κόσμο όσον αφορά την ενέργεια στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε ότι δεν εκμεταλλευόμαστε ακόμα. Αλλά και εδώ τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Είναι καλό να σκεφτόμαστε τις επιχειρήσεις μας και πώς θα προχωρήσουν. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα στην Ευρώπη από ό,τι είναι στους ανταγωνιστές μας. Από την άλλη μεριά όμως δεν εκμεταλλευόμαστε ακόμα αρκετά τις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα τον οικοδομικό 40% της ενεργειακής κατανάλωσης. Με δύο προτεραιότητες κατά τη γνώμη μου. Την μόνωση των υπαρχόντων κτηρίων και τη θέρμαση. Δεύτερον, μεταφορές, αυτός ο δεύτερος τομέας, που και εδώ πρέπει να έχει μεγάλη προτεραιότητα, η βελτίωση των κινητήρων καύσεως για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, χρησιμοποιώντας τα πιο προηγμένα υλικά για την κατασκευή των οχημάτων και κατά τη γνώμη μου τεχνολογικά σήμερα μπορούμε να περάσουμε από τα 6 λίτρα τα 100 που ισχύει σήμερα μπορούμε να περάσουμε στα 3. Δεύτερον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το ηλεκτρικό όχημα στις πόλεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Το άλλο θέμα είναι οι ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε τα μέσα να παράγουμε ηλεκτρικό εξοπλισμό που να είναι στην πρώτη γραμμή, με τις καλύτερες δυνατόν προδιαγραφές. Ένας άλλος άξονας είναι οι τιμές και το κόστος. Μόλις κάναμε μία ανάλυση που εξηγεί πολύ καλά πώς έχουν τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην χοντρική και τη λιανική τιμή. Θα πρέπει λοιπόν μαζί ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κομισιόν, κοινοβούλιο και κυβερνήσεις και διάφοροι φορείς να λάβουμε υπόψη μας τις συνέπειες. Μια άλλη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και να προχωρήσουμε περισσότερα στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Ο το τομές της ενέργειας συχνά, χωρίς με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, δεν επενδύει επαρκώς. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι δεν θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε την ανταγωνιστικότητα που θέλουμε αν μείνουμε πίσω στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στον τομέα της χρήσης των πιο προηγμένων υλικών και της πιο προηγμένης τεχνολογίας. Ένα απλό παράδειγμα. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας κοίταζα τι γίνεται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μας. την καταμέτρηση ενέργεια τους μετρητές. Φτάνουμε σε μια στιγμή που θέλουμε να διευκολύνουμε τη μαζική διανομή τους, επιτρέποντας τον καταναλωτή να καταλαβαίνει τι του γίνεται και να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση. Ε, λοιπόν, όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία για αυτού του ευφύ μετρητέ, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Συνεπώ, πρέπει να κάνουμε τεράστια προσπάθεια ακόμα για να καλύψουμε τη διαφορά και για να βρεθούμε εμείς στην πρώτη γραμμή. Και βέβαια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως όλα τα κοινοτικά κονδύλια. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζω ότι θα έχουμε 6 δισεκατομμύρια για τον ορίζοντα 2020 όσον αφορά την έρευνα. 3 δισεκατομμύρια από τα διευθυντικά ταμεία, 5,8 δισεκατομμύρια για το συνδέοντα στην Ευρώπη, Connecting Europe Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα κονδύλια να τα χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος, όπως το ακούσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, πρέπει να προσέξουμε όλους ιδιαίτερος την ασφάλεια για τα πυρηνικά πρώτα απ' όλα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τις δικές μας πρωτοβουλίες για την πυρηνική ασφάλεια, διότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ο αρχιτέκτονας της ασφάλειας αυτής. Δεν μπορεί να υπάρξουν πυρηνικές καταστροφές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν και αυτό θα το πετύχουμε συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστώ για αυτή τη γενική επισκόπηση που μας δώσατε των ε, ενεργειακών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε ακόμα στην απαρχή αυτής της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σημαντικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο μέλλον. Αλλά, όπως το τονίσατε και εσείς στην ε, αρχική σας ε, εισαγωγή, έχουμε διάφορους ομιλητές. Ξεκινώ με την κυρία Γκροστέθ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ριστόρη, λοιπόν, γιατί μας έχει παρουσιάσει ένα γενικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλήρες και μας έχει παρουσιάσει την κατάσταση της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν με αφορμή αυτά που έγιναν στην Ουκρανία και την ε, Κρυμαία βλέπουμε πόσο ουσιαστική είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο πρέπει να εργαστούμε για να το πετύχουμε αυτό και πιστεύω ότι η επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι κομβική. Θα είναι μια θητεία όπου η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση όλων των προσπάθειών μας γιατί θα έχει πολλές ε, επιπτώσεις και σε επίπεδο πολιτικής έρευνας και σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πλήρη εικόνα που μας έχετε δώσει. Θέλω να τονίσω τώρα ιδιαίτερα το θέμα του τιμήματος της ενέργειας. Τονίσατε πάρα πολύ το θέμα του κόστους της ενέργειας που πολλές φορές είναι πιο υψηλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι σε άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Είδαμε τώρα στις ΗΠΑ πόσο κατέρευσαν οι τιμές της ε, ε <clears throat> ενέργειας με την επανάσταση της χρήσης του αερίου από συστολιτικούς σχηματισμούς. Βλέπουμε τώρα πόσο αυτό επηρεάζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και βλέπουμε τον τεράστιο αυτό κίνδυνο, όπως υπογράμμισαν πολλοί, της μετακίνησης των επιχειρήσεων της λεγόμενης διαρροής άνθρακος. Και εδώ τονίζω ότι η ενεργειακή πολιτική συνδέεται άρρηκτα με τη βιομηχανική πολιτική και με το σύνολο της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει επιπτώσεις και στην πολιτική για την κλιματική αλλαγή, αλλά όχι μονάχα αυτή. Κυρίως η μεγάλη σύνδεση είναι με τη βιομηχανική πολιτική. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι την τελευταία θητεία της η Κομισιόν μίλησε πάρα πολλές φορές για την ενεργειακή πολιτική υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά χωρίς να λάβει υπόψη το μέλλον της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παραγωγή στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της ενέργειας δεν πρέπει να είναι τροχοπέδι για κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα νέο <clears throat> σχέδιο για τις κατευθυντήρες γραμμές σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις στον τομέα αυτό. Έχει ξεκινήσει από το τέλος Δεκεμβρίου μια δημόσια διαβούλευση. Εκφράζω λοιπόν την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει ένα σύστημα χρηματοδότησης της ενέργειας που να βασίζεται περισσότερο στους μηχανισμούς της αγοράς. Έχουμε κάποιες τεχνολογίες που είναι ήδη όριμε και οι οποίες δεν χρειάζονται πια δημόσιες επιδοτήσεις που το κόστος της το επομίζονται καταναλωτές αλλά ανησυχώ και για το γεγονός ότι γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια εξαιρέσεως για τους τομείς που είναι ηλεκτροβόροι. Με το να μειώνονται οι τομείς που είναι επιλέξιμοι και το να τεθούν οροφές στο συνολικό επίπεδο των ε, εξαιρέσεων φοβάμαι ότι θα αυξηθεί συνολικά το κόστος της ενέργειας για τέτοιου είδους ενεργοβόρες βιομηχανίες. Τέτοια κριτήρια λοιπόν πιο αυστηρά θα οδηγήσουν πολλούς τομείς σε ένα κίνδυνο μετακίνησης και θα ήθελα γι' αυτό να σας ρωτήσω κύριε Γενική Διευθυντά πώς εσείς δικαιολογείτε ένα τέτοιο μέλλον. Συμφωνώ μαζί σας για τις αποφάσεις οι οποίες ελέφθηκαν... στα πλαίσια της κλιματικής αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές και πραγματιστές και εντυπωσιάζομαι που θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο καθεστώς για βιομηχανίες που έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και ανάγκες ενέργειας χωρίς να λάβουμε υπόψη τις πραγματικότητες ανατομής. Για παράδειγμα, η χαλιβουργία. Έχουν πληγεί πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία, γιατί είναι μια χαλιβουργία που βρίσκεται κοντά στη βιομηχανία μας. Θα πρέπει να τη διατηρήσουμε. Είναι και η βάση ραχοκοκαλιά της βιομηχανικής πολιτικής. Πώς μπορούμε να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς χαλιβουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μιλάμε με τις κύριες βιομηχανίες μας βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα μείωσης ε, εκπομπών μέχρι το 2015, εμείς λέμε ότι μπορεί να γίνει μια μείωση 15% μοναχα και όχι 80% που ζητάει η Κομισιόν. Ίσως θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες, αλλά θα πρέπει να σταματά να αυξάνεται με τεχνητούς τρόπους η τιμή της ενέργειας, γιατί αυτό οδηγεί σε πάρα πολλούς σοβαρούς κινδύνους για τη βιομηχανία μας και για κάποιους τομείς συγκεκριμένους. Πώς μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε αυτή τη σύνδεση μεταξύ της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας ορισμένων τομέων που είναι οι ηλεκτροβόρη και φυσικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και να τη συνδυάσετε με την ανάγκη να έχουμε μια πραγματική πολιτική ενεργειακή ανεξαρτησίας. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω, μάλλον λέει ο κύριος Ριστόρη, την κυρία Γκροστέτ για το σύνολο των θέσεών της και για τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και η επόμενη κοινοβουλευτική περίοδος. Συμφωνώ επίσης και τον συσχετισμό ενεργειακής πολιτικής και βιομηχανικής πολιτικής. Έχουμε ανάγκη από μια βιομηχανική βάση στην Ευρώπη και χαίρομαι γιατί τώρα πλέον αυτό το πιστεύουν όλα τα κράτη-μέλη. Εκπλήσωμαι όταν πηγαίνω στις διάφορες πρωτεύουσε, βλέπω ότι το θέμα της βιομηχανίας είναι υψηλά. Και να σας πω ότι αυτό είναι κάτι το καινοτόμο. Δεν υπήρχε μια τέτοια αίσθηση στις διάφορες πρωτεύουσε και μας δίδει κάποιες ελπίδες ε, για το μέλλον. Σχετικά τώρα με το κόστος, νομίζω ότι η ανάλυση μας έδειξε τις διαφορές ανάμεσα στις χονδρικές τιμές και στις λιανικές τιμές. Οι λιανικές τιμές χαρακτηρίζονται από, μια, από ένα άθροισμα, αν θέλετε, επιμέρους αναλυτικών συνιστοσών, επιμέρους τιμών. Και θα πρέπει με τις κυβερνήσεις της κάθε χώρας αυτό το θέμα να το εξετάσουμε. Ε, πάντως ε, μένω και σε αυτό που είπατε στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές επιδοτήσεις για το περιβάλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια συμβατότητα καλύτερη από αυτή που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ε, στους διαφορετικούς τομείς ανάμεσα σε αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της πολιτικής του ανταγωνισμού, σεβόμενοι φυσικά τις αρμοδιότητες του καθενός και σε αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, της βιομηχανικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής. Να πω εδώ ότι τα μηνύματά μας ε, από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού περνούν γιατί υπάρχει καθήκον και υποχρέωση από πλευράς μας να δώσουμε ορισμένες εξηγήσει, να τεκμηριώσουμε τις γνώσεις μας ε, δεν είμαστε βέβαια στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής πάντα αρμόδιοι και γι' αυτό πρέπει να διευκρινίζουμε συχνά κάποιες καταστάσεις. Ιδιαίτερα σχετικά με τα κριτήρια απόκλησης για τις εντατικές χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ε, υπήρξε μια δημοσία διαβούλευση όπως γνωρίζετε ε, ε, συνεχίζεται μια δραστήρια συζήτηση ε, όπως συνηθίζεται άλλωστε πριν από τη λήψη σημαντικών υποφάσεων και ακριβώς η συζήτηση γίνεται και ανάμεσα στις διάφορες κυβερνήσεις, την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκομένους. Φτάνουμε λοιπόν σε μια απόφαση γύρω από την περίπτωση αυτή της εντατικής κατανάλωσης ενέργειας και έχει σημασία να λάβουμε υπόψη μας το σύνολο των σημείων τα οποία θέσατε και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σήμερα η αμοιβαία κατανόηση είναι υψηλότερη από ό,τι πριν μερικούς μήνες και αυτό χάρη στο σύνολο των θεμάτων των στοιχείων που μας ενημέρωσαν και από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Ε, μια συνεχής ενημέρωση δεν περνά ημέρα χωρίς να συζητάμε τα θέματα αυτά μαζί τους. Ελπίζω λοιπόν ότι πέραν του ότι τώρα υπάρχει ένα καινούριο άνοιγμα θα έλεγα προς την κατεύθυνση αυτή και από πλευράς του αρμοδίου επιτρόπου του κυρίου Αλμούνια Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουν όλοι να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο. Ο κατάλογος δηλαδή να μην είναι περιοριστικός αλλά να καλύπτει τομεακά το μέγιστο δυνατό έδαφος. Αναφερθήκατε στο αλουμίνιο, στις τσιμεντοποιίες, στο χάλιβα, στη χαρτοποιία, στη χημεία. Πρόκειται για βασικές βιομηχανικές δραστηριότητες πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη και για την ευρωπαϊκή παραγωγική βάση και για ό,τι προσφέρουν στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Σήμερα προτείνεται ένας νέος στόχος 20% του ΑΕΠ για τη βιομηχανία. Έχει χάσει πάρα πολύ ποσοστό. Χώρες ε, πριν 10 χρόνια έφτανε στο 34%. Ε, και σήμερα έχει πέσει στο 14, έχασε 20% της σημασίας της σε σχέση με το σύνολο ΑΕΠ. Απαιτείται λοιπόν η πολιτική μας να ανταλαμβάνει όλα αυτά υπόψη. Θα κρυθούμε εκ του αποτελέσματος. Πάντως πρέπει να είμαστε νομίζω κάπως πιο αισιόδοξοι σήμερα από ό,τι χθε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Ο κύριος Κορέα Δεκάμπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Διευθυντά. Αγαπητέ φίλε, θέλω να σας συγχαρώ για τον πρόσφατο διορισμό σας και είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε ένα εξαιρετικό έργο ξέροντας τι είχατε κάνει στο παρελθόν και σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σας. Έχω λοιπόν μεγάλη εμπιστοσύνη στην ε, δυνατότητα να έχουμε μια γενική διευθυνσή ενέργειας η οποία θα είναι δυναμική και η οποία θα μπορέσει να έχει ένα πάρα πολύ ενεργό χαρακτήρα μέσα στην Κομισιόν. Όλοι ανησυχούμε ιδιαίτερα για το θέμα των τιμών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως τη, την τιμή του, του βιομηχανικού ρεύματος που έχει διαφορετικό βέβαια επίπεδο σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συνολικά αν το δούμε δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις ΗΠΑ και την Κίνα ή άλλες μεγάλες οικονομικές οντότητες. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα όχι μονάχα για τον καταναλωτή αλλά και για τις βιομηχανίες. Υπάρχει μεγάλη ψαλίδα μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής <clears throat> ενέργειας και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αρχίζει να φαίνεται στα λεγόμενα ευφυή δίκτυα για τον καταναλωτή. Έχουμε να αποθέσει πάρα πολλές ε, ελπίδες στα λεγόμενα εφηδίκτια για τους καταναλωτές και βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νομίζαμε να γίνει ο καταναλωτής καλός διαχειριστής της κατανάλωσης ενέργειάς του. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά προβλήματα. Συμφωνούμε όλοι με την ενισχυμένη περιφερειακή προσέγγιση σας για, την, ε, για τις διασυνδέσεις και συμφωνούμε όλοι για τον ίσονα χαρακτήρα, για τον αμεληταίο σχεδόν χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επιτυχία των ε, διασυνδέσεων. Εμείς είδαμε ότι ο στόχος του 10% και είναι πολλές οι χώρες οι οποίες δείχνουν δυσαρέσκεια με όλα αυτά που έχουν γίνει σε επίπεδο διασυνδέσεων. Υπήρχε μια πρωτοβουλία 11 χωρών μελών, μεταξύ των οποίων και η Πορτογαλία, για να επιτευχθεί ένας στόχος πιο φιλόδοξος από αυτόν που είχαμε στο παρελθόν. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα στόχο 30% βελτίωση σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια ήταν η, αντίδραση της Κομισιόν για τις προτάσεις αυτές. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η επίσημη πρόταση της Κομισιόν. 40% αύξηση της αποδοτικότητας και υπάρχει φυσικά η, αλλαγή ε, διατύπωσης από αποτελεσματικότητα σε αποδοτικότητα. Είναι ασαφής αρκετά ο στόχος του 30% μέσα σε κάθε κράτος μέλος και το 40% ενεργειακής αποδοτικότητας είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά αλλά είναι πάνω επιπλέον αυτών που έχουν επιτευχθεί ε, από το 1990 μέχρι τώρα. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν πάρα πολύ φιλόδοξα, αλλά δεν είναι. Χαιρόμαστε λοιπόν που είστε ενώπιόν μας και μπορούμε να βασιζόμαστε στη δική σας βοήθεια για τον ορίζοντα 2020 σε ό,τι αφορά τα θέματα των διασυνδέσεων την έρευνα και την τεχνολογία, τα 3 δισεκατομμύρια για τα περιφερειακά θέματα. Όλα αυτά όμως παραμένουν ακόμα σε ένα επίπεδο ασάφειας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να γνωρίζω και πιστεύω όλοι μας είναι ποια ακριβώς είναι η θέση της Κομισιόν και της Γενικής Διευθύνσεώς σας σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους του, της εξοικονόμησης 30% χάρη στις καλύτερες διασυνδέσεις. Αν δεν λύσουμε αυτά τα προβλήματα, δεν θα φτάσουμε ποτέ σε μια κοινή αγορά ηλεκτρισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον μια διαπεριφερειακή αγορά ηλεκτρισμού. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τρεις συναδέρφους. Ήβαν... Και μετά τους τρεις συναδέρφους θα απαντήσει ο κύριος Ζήστορη. Ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο πρώτα απ' όλα. Καταρχάς ξεκινώντας θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ευθύνη την οποία έχετε αναλάβει στον τομέα της ενέργειας, κάτι το απόλυτα κομβικό στις περαιτέρω πολιτικές μας. Θα ήθελα να προσπαθούσουμε να δούμε μια διαφορετική εφαρμογή των προβλέψεων της ενεργειακής πολιτικής με πιο συστηματικό τρόπο παρούσης και στις υπόλοιπες πολιτικές. Θα πρέπει δηλαδή έτσι η ενέργεια να βοηθήσει και τους υπόλοιπους τομείς. Φέρνω εδώ σαν παράδειγμα το θέμα της βιομάζας και τα υπόλοιπα δασικά και ε, αγροτικά απόβλητα ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μολυσμένες περιοχές για την ε, βελτίωση του εδάφους και θα μπορούσαν επίσης να γίνουν αντικείμενο πυρολιτικής επεξεργασίας για παραγωγή υδρογόνου. Ε, Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε τόνος ξηράς βιομάζας μπορεί να παράγει ε, χίλια κυβικά μέτρα υδρογόνου και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε θα έλεγα αυτό το καύσιμο και θα έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε και τις ε, αναφλέξεις που δημιουργούν προβλήματα μόλυνσης στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα δημιουργίας με συστηματικό τρόπο παραγωγής ενέργειας σε σχέση με την προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το έδαφος με πολύ λεπτομερή και παρεμβατικό τρόπο. Κάτι τέτοιο αν δεν το κάνουμε δεν θα εκμεταλλευτούμε σωστά την ενέργεια η οποία μας προσφέρεται. Μαζί λοιπόν με την δυνατότητα αποφυγής της ανάφλιξης. Ε, ένα άλλο θέμα είναι αυτό το οποίο έχει αρχίσει να έρχεται στην επικαιρότητα με τα μεγάλα αιωλικά offshore πάρκα στη θάλασσα δηλαδή. Πράγματι αυτά τα πεδία τα αιωλικά έχουν την δυνατότητα απορρόφησης ενός μεγάλου τμήματος της ενέργειας των καταιγίδων. Αυτό ε, μπορεί να φτάσει το 1 τρίτο περίπου της ισχύω τους και αυτό μπορεί να βελτιώσει τις κλιματολογικές συνέπειες σε κάποιες ε, ε, παράκτιες περιοχές που φύγονται από τέτοιου είδους θαλάσσιες καταιγίδες και νομίζω ότι αυτές οι θαλάσσιες αιωλικές εγκαταστάσεις θα προσφέρουν πολλά. Όλα αυτά λοιπόν θεωρώ ότι μπορούν με πιο συστηματικό τρόπο να γίνουν πραγματικότητα και να δημιουργήσουμε έτσι μια μεγαλύτερη εναργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης ε, και να βοηθήσουμε και πολλούς άλλους τομείς. Έχει ακουστεί πολλές φορές αυτό που θα πω, αλλά είναι σαφές ότι το να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ηλεκτρικό υψηλής αποδοτικότητας, υψηλής τάσης και κυρίως συνεχούς τάσης είναι κάτι το απαραίτητο για την βέλτιστη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμα και ο άνθρακας που δεν είναι ανανεώσιμος μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πυρόληση και να αποφύγουμε έτσι την ανάφλεξή του και τις περιβαλλοντικές συνέπειες που έχει. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία έτσι ώστε να ικανοποιηθεί από τη μία η ανάγκη που έχουμε σε ενέργεια και από την άλλη να δώσουμε περισσότερες εγγυήσει για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βινταλ Κουάντρας τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια αγαπητέ κύριε Ριστορή, που διοριστήκατε γενικός ε, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας. Νομίζω ότι το βιογραφικό σας ε, προφανώς και σας οδηγεί σε αυτή τη θέση. Είσαστε στην θέση την πιο κατάλληλη για σας. Ήταν ο προορισμός σας. Ξέρετε όμως από την άλλη μεριά ότι όταν κανείς δημιουργεί πολλές προσδοκίες ε, πρέπει μετά να αντέξει. Είμαστε όμως σίγουροι ότι θα τα καταφέρετε. Διαπιστώσαμε στην παρέμβασή σας ότι μας και γραφίσατε ένα, μια πλήρη εικόνα της ενεργειακής μας πολιτικής, έτσι πολύ γρήγορα, με την ικανότητά σας να συνθέτετε στα διάφορα θέματα. Μας μιλήσατε χωρίς κανένα κόμπλεξ για την ανταγωνιστικότητα και για το πώς θα ισορροπήσουμε την ανταγωνιστικότητα με την βιωσιμότητα. Είπατε ότι πρέπει να καταργηθούν επιδοτήσεις για τις τεχνολογίες που φτάνουν σε κάποιο βαθμό ρημότητας. Υπογραμμίσατε επίσης ότι υπάρχουν χώρες που δεν είναι ανταγωνιστικές ενεργειακά και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και μας υπενθυμίσατε επίσης ότι το ενεργειακό μείγμα πρέπει να είναι ισορροπημένο, διαφοροποιημένο χωρίς δογματικές προκαταλήψεις για τη μία την άλλη μορφή ενέργειας. Όλα αυτά πολύ καλά. Είναι λόγια αυτά που βρίσκουν πολλούς από εμά σύμφωνους και που ευχάριστα τα ακούμε. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, για την αποτελεσματικότητα, τις εναλλακτικέ ενέργειες και τους στόχους. Για ποιο λόγο επιμένουμε ακόμα σε δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τις εναλλακτικέ ε, ενέργειες, κάτι που είναι αρνητικό για την αποτελεσματικότητα. Ξέρω ότι εσείς αυτό το κληρονομήσατε βέβαια από τους προκατόχους σας, αλλά θα έπρεπε επιτέλους, μια και έξω, να τολμήσουμε να πούμε ότι η αποτελεσματικότητα πρέπει να μπει στο ίδιο επίπεδο να και την ίδια στρατηγική σημασία με τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με την χρηματοδότηση. Όλο όσα είπατε είναι αλήθεια. Οι διασυνδέσεις, νέες τεχνολογίες, βελτίωση προδιαγραφών, καθαρή τεχνολογία άνθρακα, ηλεκτρικά οχήματα. Ο κύριος Πρόντι μας υπενθύμησε και άλλα για το υδρογόνο. Οι ανάγκες μας τα επόμενα χρόνια, ανάγκες ανανέωσης των εγκαταστάσεών μας, παραγωγής ενέργειας είναι πράγματα τα οποία απαιτούν τεράστια χρηματοδότηση. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια. Πώς λοιπόν θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πού θα τα βρούμε τα χρήματα αυτά. Αυτό το τεράστιο όγκο επενδύσεων που χρειαζόμαστε. Και αυτό για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία εσείς αναφέρατε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ριστόρη, κύριε Γενικέ Διευθυντά και συγχαρητήρια για το διορισμό σας. Θέλω να σας ρωτήσω για το ξεκίνημα και για την εφαρμογή του ορίζοντα 2020. Ξέρετε, εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μεγάλε φιλοδοξίε. Αυξήσαμε βασικά και τι φιλοδοξίε και το εύρο εφαρμογή και τον προπολογισμό. Ομόφωνα μάλιστα. έχουμε υπογραμμίσει έχουμε υπογραμμίσει όλος ιδιαιτέρως το θέμα της ευφύους ενέργειας για την Ευρώπη. Είναι καλό που μπήκε στον ορίζοντα 2020 γιατί έτσι υπάρχει μια συνέχεια στις δραστηριότητες. Και επίσης υπογραμμίσαμε πολύ στις βιομηχανικές εφαρμογές. Πιστεύουμε ότι κάποιες τεχνολογίες έχουν φτάσει σε επίπεδο οριμότητας, οπότε τώρα αυτό που χρειάζεται είναι εφαρμογή σε, σε μεγάλη κλίμακα. Η έρευνα, η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας ε, σήμερα για να καλυφθεί το τρίγωνο αυτό που έχει να κάνει με την ενέργεια, την αποτελεσματικότητα και προκειμένου να μπορούμε να έχουμε τεχνολογίες που να είναι και πιο καθαρές και να κοστίζουν λιγότερο και να έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Συνεπώς, θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσείς πώς βλέπετε να εφαρμόζονται όλα αυτά ποια θα είναι η σχέση με τις άλλες γενικές διευθύνσεις που εφαρμόζουν τον ορίζοντα 2020. Βλέπετε εσείς να υπάρχει μια εξέλιξη στις σχέσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κ. Μασέκεβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ριστόρη για τον πρόσφατο διορισμό του ως Γενικό Διευθυντή. Έρχομαι από την Πολωνία, όπως ξέρετε, μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Και πρέπει να πω ότι ξεκίνησαν πολύ καλά με την έκθεση Βιντάλ Κουάδρας. Αλλά στην Ουκρανία, ήταν τότε που μάλλον στην Ουκρανία είχαν κλείσει τις τρόφιγγες οι με σημαντικές επιπτώσεις. Τότε συντάξαμε ένα κανονισμό που ετέθη σε εφαρμογή με την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Τώρα έχουν περάσει κάποια χρόνια, είμαστε στο 2014 και πάλι έχουμε ενώπιόν μας το πρόβλημα της Ουκρανίας και βλέπουμε ότι η κοινότητα ενέργειας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες. Είμαστε πάρα πολύ πολύμορφοι μεταξύ του Βορρά, μεταξύ του Νότου, της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης. Κάθε περιοχή στην Ευρώπη, κάθε περιφερειακή οντότητα έχει διαφορετικό επίπεδο βιομηχανίας και επίσης έχει διαφορετικές μορφές παραγωγής ενέργειας που έχουν φυσικά διαφορετική ιστορία. Έχουν δημιουργηθεί μέσα σε δεκαετίες στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι που έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Με την ε, επιβολή στόχων για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την κυρία Κροστέτ, ήταν ατυχής αυτή η επιζήτηση λύσης επί τη βάση μοναχά της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι τώρα είχε αντιμετωπίσει υπερβολικά από το πρίσμα της μέσα από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας τα ενεργειακά θέματα. Χρειαζόμαστε πιο στιβαρή αντιμετώπιση από εσά από τη δική σας Γενική Διεύθυνση, α, γιατί ακόμα από την Κομισιόν δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι. Οι πράσινοι στόχοι που είχαν τεθεί δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τις ανάγκες της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Μιλούσαν κάποιοι για ενεργοβόρες βιομηχανίες. Μα αυτές οι ενεργοβόρες βιομηχανίες είναι που δίνουν θέσεις απασχολήσεως και εκεί είναι και το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί θέτουμε φιλόδοξους στόχους που είναι ανέφικτοι. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενότητα για τα θέματα ενέργειας. Και θέλω να θέσω και ένα σύντομο ερώτημα, εάν μου επιτρέπετε για την ε, συνεδρία του Συμβουλίου που θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Σίγουρα θα υπάρξουν συζητήσεις για τα θέματα αυτά που προανέφερα. Το ερώτημά μου προς εσάς είναι αν θεωρείτε ότι είναι πιθανό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ενεργειακούς μας στόχους από ένα διαφορετικό χώρο και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, και ανεξάρτητη από τον Πούτιν. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Χιούμπνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πρέπει να αποδεχτώ, ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο όταν σας βλέπω να αναλαμβάνετε αυτό το αξίωμα. Συγχαρητήρια λοιπόν και από μένα και είμαι πιο αισιόδοξη τώρα για την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη. η ενέργεια είναι το α και το ω της βιομηχανίας στην Πολωνία. Χωρίς ενέργεια, χωρίς το σωστό ενεργειακό μείγμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αν δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την εξάρτηση από τρίτες χώρες που μας παρέχουν ενεργειακούς πόρους, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Θα φύγει η βιομηχανία από την Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας έχει ήδη φύγει. Όλα αυτά που λέτε λοιπόν είναι πολύ σωστά. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να δούμε. Μιλήσατε για την καινοτομία παραδείγματος χάρη. Τα νέα μέτρα για την συγκράτηση και ε, αποθήκευση άνθρακος είναι απαράδεκτα. Αυτά που γίνονται για την πυρηνική ενέργεια δεν είναι αποδεκτά. Η βιομάζα δεν μας έχει βοηθήσει παρά μόνο περιορισμένα γιατί μειώνει και την αγροτική παραγωγή. Και το ερώτημα είναι με τον άνθρακα, τι θέλουμε να κάνουμε με τον άνθρακα και πώς θα λειτουργήσουν οι ανανεώσιμες ενέργειες όταν είναι τόσο ψηλές και δεν είναι υψηλότερε μόνο γιατί επιδοτούνται οι ανανεώσιμες ενέργειες. Δεν έχουμε λοιπόν ακόμα τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Προς τα πού λοιπόν θέλουμε να κινηθούμε. Μιλήσατε για διπλώματα τεχνίας, για καινοτομία λέτε ότι εμείς υπολοιπόμεθα πίσω από, την, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και από την Κίνα. Αλλά αυτές οι διαδικασίες καινοτομία χρειάζονται πολύ χρόνο. Εγώ θα έκανα οτιδήποτε είναι δυνατό για να μειωθεί αυτός ο χρόνος υστέρησης. Κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι για να θεσπιστούν προτεραιότητες στους τομείς αυτούς. Και πώς, κύριε Γενική Διευθυντά, θα εξασφαλίσετε ότι το ενεργειακό μείγμα στην Ευρώπη δεν αποκλείει ορισμένο οποιαδήποτε πηγή και πώς θα εμποδίσετε την διαρροή των επιχειρήσεων προς άλλες περιοχές του κόσμου. Πού θα μας φέρετε σε αυτό το σημείο, με ποιο δρόμο, με ποια κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε μονάχα μία ατελή αγορά ανανεώσιμης ενέργειας. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να βρούμε μια πραγματική λύση αν δεν αφήνουμε τις άλλες μορφές ενέργειας να ανθίσουν. Ευχαριστώ λέει Τελευταία ερώτηση. Έχετε το λόγο πάλι κύριε Ριστορή γιατί πράγματι τα θέματα αυτά παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθμό δυσκολίας και περιπλοκότητας. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που πήραν το λόγο. Θέλω να απαντήσω καταρχάς στον κύριο Κορέντε Κάμπος σχετικά με τις τιμές. Έχουμε ήδη παρουσιάσει μία ανάλυση, για πρώτη φορά θα έλεγα τόσο πραγματικά λεπτομερή. Από την ανάλυση αυτή <clears throat> θα έλεγα μπορεί κανείς να καταλήξει σε ορισμένες διαγνώσεις και τις πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χονδρικές τιμές και στις λιανικές τιμές στις χονδρικές τιμές οι τιμές του φυσικού αερίου είναι σταθερές και οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι οι χαμηλότερες τα τελευταία 10 χρόνια. Συγκρίσιμες πλέον με τις αμερικανικές τιμές που είναι χαμηλές. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με αυτό, κυρίως μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν ανάμεσα σε διάφορες πλευρές της ενεργειακής πολιτικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. Πολλές χώρες θεώρησαν ότι πρέπει να μεταφέρουν στους καταναλωτές ε, και τα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες το βάρος των επιδοτήσεων που στην ουσία δημιουργούν όχι μόνο στρεβλέψεις του ανταγωνισμού αλλά και περισσότερα προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι την πληρώνουν λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα θα πρέπει να ήταν πρωταγωνιστές της βιομηχανικής βάσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη και να προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά χρήζουν προστασίας. Και σας θυμίζω ότι σε επίπεδο τιμών η κατάσταση διαφοροποιείται κατά πολύ από τη μία χώρα στην άλλη και στον τομέα των τιμών για τη βιομηχανία και στον τομέα των ε, τιμών για τα νοικοκυριά. Κάποιες κυβερνήσεις ε, ε, επέτρεψαν να υπάρξουν αποκλήσεις για τη βιομηχανία και άλλες κυβερνήσεις οι οποίες έπαιξαν με μορφές προστασίας για το κόστος του ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε εδώ σε όλα αυτά πιο, ε, πιο δημοκρατικά και πιο ευρωπαϊκά. Τώρα έχουμε στα λεγόμενα FEE e δίκτυα και το κομμάτι που αφορά τον καταναλωτή. Σύμφωνο μαζί σας και το είπα στην παρέμβασή μου, στην εισαγωγή μου. Ανησυχώ για την καθυστέρηση που σημειώνει η Ευρώπη στον τομέα της έρευνας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τους e και μέτρητες κτλ δηλαδή τις δυνατότητες που έχουμε να δώσουμε στον τελικό καταναλωτή τον σωστό έλεγχο της κατανάλωσής του και την παρακολούθηση του κόστους της κατανάλωσής του. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό σήμερα να είμαστε τόσο πίσω όχι μόνο από τους Αμερικανούς αλλά και από τους Ασιάτες και τις κινέζικες επιχειρήσεις. Σας θυμίζω ότι το μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης είναι η ιδιωτική κατανάλωση και ακολουθείται από τις βιομηχανίες. Και θέλω λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμφωνήσουν έτσι ώστε να ανακάμψουμε διότι δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε μείνει τόσο πίσω σε τομείς καθοριστικούς για το μέλλον μας. Πρέπει λοιπόν ε, να σημειώσουμε πρόοδο γενικότερα στα ICT και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω του μείωσης του κόστους της ενέργειας. Για τις διασυνδέσεις συμφωνώ με αυτά που είπατε. Εύχομαι και εγώ να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε λίγο στο θέμα και να καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένα δεδομένα και αριθμούς για την πρόοδο που έχει συντελεστεί, για την πρόοδο που δεν έχει συντελεστεί ε, και ιδιαίτερα για τις πιο ευαίσθητες ε, περιοχές και θέλω να επανέλθω και εδώ και προς το Συμβούλιο με πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Θα πρέπει παράλληλα να σας πω ότι έχοντας συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τους υπευθύνους των Ισπανικών και Γαλλικών δικτύων, πράγματι κάποια σημαντικά βήματα προόδου έχουν γίνει σε τομείς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί σαν δύσκολοι και υψηλού κόστους και τεχνολογικά απαιτητικούς. Πρέπει λοιπόν να επαναξιολογηθεί η κατάσταση και επί τη βάση αυτής της επαναξιολόγησης να επανέλθουμε με αυξημένες αυτή τη φορά φιλοδοξίες γιατί μεσοπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε και να προβλέψουμε τη σωστή πορεία των ευρωπαϊκών αγορών προβλέποντας πάντα βέβαια και βελτιώσεις σε επίπεδο περιφερειακό. Ο κύριος Πρόντι έχει δίκιο όταν αναφέρεται στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τη βιομάζα και γύρω από τα αγροτικά και δασικά απόβλητα. Αναφέρθηκε στην πυρόληση για την παραγωγή του υδρογόνου. Φυσικά έχει ενδιαφέρον αυτό και θα πρέπει όλες αυτές τις επιλογές να τις λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε εμείς να στερήσουμε τον εαυτό μας από αυτού του είδους τους ενεργειακούς πόρους. Και σωστό είναι αυτό που είπατε και για τα αιωλικά πάρκα στη θάλασσα. Εκεί έχουμε πραγματικά μείνει πάρα πολύ πίσω. Θα πρέπει να διακρίνουμε βέβαια το τι έχει ήδη οριμάσει μέχρι τώρα, δηλαδή τα πάρκα, τα φωτοβολταϊκά και το αιωλικά, ε, σε ε, στερεό έδαφος. Έχετε δει ότι έχουμε γίνει εδώ σχετικά ανταγωνιστικοί όπως επίσης και τα μεγάλα αιωλικά πάρκα offshore που είναι ένα τεχνολογικό, ε, μια τεχνολογική πρόκληση τεράστια και έχει σχετικά υψηλό κόστος ακόμα αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δοκιμαστεί και για τον λόγο για τον οποίο είπατε, δηλαδή τη μείωση των βίαιων κλιματολογικών φαινομένων όπως τα τσουνάμι και οι καταιγίδε που φύγουν τις παράκτιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που είπατε για τον άνθρακα και την πυρόληση και τα δίκτυα υψηλής αποδοτικότητας και αυτά είναι προκλήσεις σημαντικότατες γιατί θα επιτρέψουν να μειώσουμε το κόστος και να μειώσουμε και τις απώλειες ενέργειας στα δίκτυά μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και τα ICT έτσι ώστε να μεταφέρουμε σωστά και γρήγορα την ενέργεια και μου κάνει εντύπωση αρνητική η έλλειψη δυνατοτήτων των εταιριών να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες μερικές φορές. Πρέπει να το κάνουν για να προχωρήσουμε με ταχύτητα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τον Βιντάλ Κουάντρας τώρα. Θέσατε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πράγματι θα πρέπει να υπάρξει ένα σωστό επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας, το ίδιο και για τις παραδοσιακές πηγές και τις εναλλακτικές. Θα κάνουμε προτάσεις μετά το καλοκαίρι. Θα αξιολογήσουμε καταρχάς το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι πρώτοι υπολογισμοί δείχνουν πως πηγαίνουμε σε μία διαφορά 17% ή μάλλον σε ένα στόχο 17% ε, και όχι 20% το 2020 έχει υπάρξει πρόοδο στην αποδοτικότητα, την ένταση μάλλον στον τομέα τον ενεργειακό και πρέπει να συγχαρούμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε όμως περισσότερες δυνατότητες που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στις κατοικίες, στις μεταφορές και γενικότερα στους εξοπλισμούς. Και πρέπει εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Για τη δεύτερη ερώτησή σας, πράγματι έχουμε ανάγκες ε, κολοσιαίες, ανάγκες ε, χρηματοδότησης. Φτάνουν αυτή τη στιγμή 500 δις. 500 δις. Και θυμίζω ότι πάρα πολλές μονάδες ε, παραγωγής, πυρηνικές ή φυσικού αερίου και άνθρακα τερματίζουν την ζωή τους την επόμενη δεκαετία. Λοιπόν, 500 δις πρέπει να επενδυθούν στον τομέα αυτό μέχρι το 2030. Υπάρχει επίσης το θέμα της μεταφοράς και διανομής που είναι άλλα 600 δις μέχρι το 2035. Γιατί θυμίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το δίκτυο που έχει αυτή τη στιγμή φτάσει σε κατάσταση γύρατος και δεν έχει προγραμματιστεί για την περιφερικότητα και την ένταση που χαρακτηρίζει τα σημερινά δίκτυα. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε τις ανταλλαγές ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από καλές συνθήκες, τη χρήση και ένταξη ε, των ε, αναλλακτικών πηγών ενέργειας και ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. 20% εναλλακτικές πηγές για την ηλεκτρική ενέργεια σήμερα. Θα πρέπει όμως να θέσουμε το θέμα αυτό και μακροπρόθεσμα. Γιατί τις θέτουμε πολλές φορές όπως τις θέταμε όταν οι εναλλακτικές πηγές δεν ήταν παραπεριθωριακές. Ζήτηση και αποθήκευση επίσης. Η αποθήκευση δεν ήταν προτεραιότητα τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να καταστεί προτεραιότητα όχι μόνο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αλλά και για τον ηλεκτρισμό. Γνωρίζετε, κάποιοι από εσά άλλαστε ήταν ιδιαίτερα στρατευμένοι στα θέματα της έρευνας. Έχουμε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας αφορά την υδρόλυση, ε, σταθερά επίπεδα <coughs> αποθήκευσης και δεύτερον τα κτίρια. Θα πρέπει να οργανώσουμε έτσι τα πράγματα για να υπάρξει για τους ισορευτές μια ευρωπαϊκή πραγματικά απάντηση. Τώρα για την απόσβεση των επενδύσεων. Για την ενέργεια έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο από άλλους τομείς που απαιτούν και αυτοί οι επενδύσεις και αναφέρομαι στις μεγάλες μεταφορικές υποδομές. Έχουμε λοιπόν καταρχάς ανάγκη από ένα σταθερό πλαίσιο έτσι ώστε να δώσουμε στις επενδυτές την προβλεψιμότητα την οποία απαιτούν. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από ένα τέτοιο πλαίσιο και δεύτερον θα πρέπει εμείς να παρουσιάσουμε τις ανάγκες μας από κοινού με τους χρήστες σε επίπεδο χρηματαγορών. Ξέρετε ότι έχουμε βιώσει μια πάρα πολύ δύσκολη από το 2008 χρηματοπιστωτική κρίση ε, τώρα αρχίζουμε να βρίσκουμε μια κάποια ρευστότητα και τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και η ενέργεια πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις επενδύσεις για την πραγματική οικονομία να κινητοποιήσουμε τις χρηματαγορές, ε, τα πιστοτικά ιδρύματα, τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία στα νομικά διασφαλισμένα πλέον πλαίσια. Από κοινού και με τη δική σας στήριξη. για την κυρία Καρβάλιο, θα ήθελα να σας πω ότι και με τον συνάδελφο Γιάν Σμίτς και τις ομάδες του συνεργαζόμαστε πλήρως για την εφαρμογή ε, της, του προγράμματος Ενέργεια 2020. Σαν παράδειγμα, εγώ προσκαλώ τακτικά τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Στρόσμεγερ, ή τον ε, αρμόδιο ε, διευθυντή έτσι ώστε να προετοιμάζουμε σωστά τα σημαντικά θέματα. Γνωρίζετε ότι θα πρέπει να επανεπικαιροποιήσουμε το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας και να το εξισορροπήσουμε με τις δικές μας προτεραιότητες, δηλαδή και με το θέμα της προσφοράς, στήριξη της ανανεώσιμες, στήριξη στα CCS, όπως επίσης να δούμε ακριβώς τι θα γίνει και με τη ζήτηση. Και εδώ τίθεται το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ξέρετε ότι έχουν υπάρξει κάποιες εμπειρίες στο παρελθόν, κάποτε πετυχημένες, κάποτε όχι. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από όλα αυτά και πρέπει να μπορέσουμε να ταξινομήσουμε τις προτεραιότητές μας και για τα ευφυή δίκτυα στο απαιτούμενο επίπεδο. Σήμερα το πρωί σε μια κοινή συνάντηση άλλωστε αποφασίσαμε να επιταχύνουμε ε, την προετοιμασία του ολοκληρωμένου οδικού χάρτη έτσι ώστε να είμαστε σε θέση μετά το καλοκαίρι να έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Ως προς αυτό, η συνεργασία ανάμεσα στις γενικές διευθύνσεις είναι λειτουργική και δεδομένη, δίδει ελπίδες για το μέλλον και τη σωστή εξισορρόπηση της ζήτησης με την προσφορά. Προς τον κύριο Βασικίβιτς, να πω ότι η κρίση με την Ουκρανία επιτρέπει καταρχάς να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό που κάναμε μετά από την κρίση του 2009. Ήδη από την αρχή της κρίσης αυτής, την Κυριακή, συνεκάλεσα εμείς, εγώ μία, μία συνάντηση της ομάδας Gas Coordination Group που συνεδρίασε τη Δευτέρα και αυτό επέτρεψε την Τρίτη στο Συμβούλιο Ενέργειας να έχουμε ακριβώς την ακριβέστατη εικόνα της κατάστασης. Την προηγούμενη Παρασκευή συνεδρίασε εκ νέου αυτή η ομάδα για να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί η κατάσταση και τη μετακόμιση ενέργειας. Ταυτόχρονα κάνουμε τα μέγιστα δυνατά για να βοηθήσουμε την Ουκρανία σε αυτή την δύσκολη μεταβατική φάση και για το σύνολο της ενέργειας. Όχι μόνο φροντίζοντας ε, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά, δηλαδή να υπάρχουν τα, οι ροές ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία και την Ουγγαρία και την Ουκρανία, χαμηλές ποσότητες βέβαια, και γι' αυτό φτιάχνουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο αν υπάρξει πολιτική στήριξη μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τον επόμενο χειμώνα και αποτελεί στην σύνδεση του αγωγού φυσικού αερίου ανάμεσα ε, στην ε, Ουκρανία και τη Σλοβακία ε, με την, με την αποθήκη φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Αυτό θα βοηθήσει κατά πολύ τη σταθεροποίηση και διασφάλιση την κατάσταση στη χώρα αυτή. Θα κάνουμε... θα ξεπεραστεί η σπάνης πόρων για τη χώρα αυτή. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Πέραν αυτών, αυτό το οποίο μπορώ να σα πω είναι ότι ο διάλογος που έχουμε με τις πολωνικές αρχές είναι μόνιμος διάλογος, ένας διάλογος ο οποίος συνεχίζεται. Και είμαστε σε επαφή με τους συμβούλους του Πρωθυπουργού του κυρίου Τούσκ. Ήμουν ο ίδιος στην Πολωνία πριν από δύο εβδομάδες και είμαι πεπισμένος μεταξύ των μέτρων τα οποία προτάθηκαν στο τέλος του Ιανουαρίου. Πολλά από αυτά πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που έχουν ε, υποστηριχθεί και από την Πολωνία. Όχι μονάχα την ε, υποστήριξη των διασυνδέσεων, αλλά και τη μεγαλύτερη ελευθερία για τα κράτη να αποφασίσουν για το μείγμα ενέργειά τους. Μια καλύτερη προσέγγιση προς την αγορά για τις ανανεώσιμες ενέργειες και επίσης και το άνοιγμα της ε, ε, αξιοποίησης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Έχουμε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση και μια σύσταση η οποία προστίθεται στην νομοθεσία η οποία ισχύει και επιτρέψει στις χώρες οι οποίες το επιθυμούν με μια ε, θεμητή από πλευράς περιβάλλοντος προσέγγιση να κάνουν διερευνήσεις για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Προσπαθούμε να αντλήσουμε λοιπόν όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα μέσα στους επόμενους 18 μήνες ή 2 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν νομίζω ότι πλησιάσουμε πάρα πολύ αυτά που ζητήθηκαν από τις αρχές της Βαρσοβίας. Και φυσικά συνεχίζουμε το διάλογο και για την άλλη πτυχή που σας ενδιαφέρει για τα αντισταθμίσματα που μπορούν να αποφασιστούν σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και που έχουν να κάνουν με τη μακροοικονομική ισορροπία στην Πολωνία. Για την κυρία Ιμπνερ, σας λέω ναι, χρειαζόμαστε μια ενεργειακή πολιτική η οποία συγχρόνως στηρίζει τη βιομηχανία μας. Η ενεργειακή πολιτική είναι σημαντικός συντελεστής για την υγεία της βιομηχανίας και εγώ ε, ετήσει και του συναδέλφου μου για από τη Γενική Διεύθυνση του Επιχείρην θα συναντήσουμε το Γενικό Διευθυντή Βιομηχανίας για να συντονίσουμε περαιτέρω τις ενέργειές μας. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία ελέγχθησαν για τι ενεργοβόρε βιομηχανίες σε ό,τι αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις. Εκεί σίγουρα η σύνδεση κλιματικής αλλαγής και ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική και ο κατάλογος των εξαιρέσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε την πολιτική μας σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες ίδιες ενέργειες για να κρατήσουμε το θετικό του χαρακτήρα, αλλά να τις κάνουμε να υπόκεινται περισσότερο στις δυνάμεις της αγοράς και αυτό είναι πολύ σημαντικό <clears throat> και σε ό,τι αφορά την αποθήκευση της ενέργειας θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα για να ανοίξουμε νέους δρόμους που δεν υπήρξαν στο παρελθόν αλλά τώρα γίνονται απαραίτητοι για να μπορέσουμε να, να επιτύχουμε τις απαραίτητες πρόοδους και στην αγορά εργασίας, στην αγορά ηλεκτρισμού και την διατήρηση των απαραίτητων διασυνδέσεων. Πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν στην Ευρώπη την ε, σύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκού επίπεδου και ευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά και εκεί οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να παραμείνουν σε σύνδεση με τα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα. Δεν είναι καλό το ότι πολλά από τα πανεπιστήμια μας είναι πολύ μακριά από τα κύρια θέματα προτεραιότητας σε σχέση με την ευρωπαϊκή βιομηχανία μόνο με κοινέ προσπάθειες όπως γίνεται ήδη στο δικό μας επίπεδο για να έχουμε καλύτερη σύνδεση μεταξύ ενεργειακής πολιτικής, βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής έρευνας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καρπού στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντά για τις πάρα πολύ λεπτομεριακές απαντήσεις που δώσατε σε όλα τα ερωτήματα των βουλευτών. Εξ ονόματος φροντός συναδέλφου μου, θέλω να σας συγχαρώ και πάλι <clears throat> για τα νέα σας καθήκοντα και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα καθήκοντα αυτά για τη δική μας Επιτροπή και είμαι σίγουρος ότι και εσείς και οι συνεργάτες σας θα είσαστε σημαντικοί εταίροι της Επιτροπής μας και φυσικά των ε, μελών που θα επανέλθουν μετά τις εκλογές. Νομίζω θα το διαπιστώσουν και αυτοί πολύ γρήγορα. Αυτοί που θα έρθουν μάλλον μετά τις εκλογές. Η Επιτροπή αυτή είναι μια Επιτροπή με υψηλή εμπειρογνωμοσύνη και για μένα ήταν τιμή να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε με την Ουκρανία, με τη μετατόπιση στις παγκόσμιες αγορές και όλα τα άλλα αστάθμητα τα οποία μπορούν να προκύψουν ελπίζω ότι θα επιτυχετε σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας και ελπίζω ότι θα ξανάρθετε στην Επιτροπή μας και θα είναι πάντα τόσο επικοδομητικές. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ συλλογικά λέει και ο κύριος Ιστόρη. Τώρα, ένα τεχνικό ζήτημα. Στις 5.30 θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών.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 Ευχαριστώ. λάβει και στις 5.30 ε, έχουμε τους συντονιστές. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν στον χρόνο. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια συζήτηση με τη Μαρία Κριστίνα Ρούσο, Διευθύντρια Διεθνούς Συνεργασίας. Την καλωσορίζουμε. Ίσως να καθυστερήσουμε λίγο τους συντονιστές. Όλοι έχετε στη διάθεσή σας ε, τα έγγραφα τα οποία έχουν διανεμηθεί προς όλους τους βουλευτές σχετικά με τη διαδικασίες των εργασ... και των ε, χρονική ε, διαδοχή. Θα δώσω το λόγο πάντως στην κυρία Ρούσο πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, εδώ στην Επιτροπή Ήτρε, όσον αφορά την διεθνή συνεργασία για την έρευνα και την καινοτομία. Τα καθήκοντά μου τα ανέλαβα τον Ιούλιο που μας πέρασε και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι υπό την ιδιότητα αυτή εδώ στην Επιτροπή σας. Θα είμαι σύντομη, γιατί όπως υπόθηκε, σας έχουμε στείλει λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τις συμφωνίες σύνδεσης. Πάντως, στην παρουσίασή μου εδώ, θέλω να σας αναφέρω τα κύρια σημαντικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, οι συμφωνίε σύνδεση αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκή Στρατηγική για συνεργασία στον τομέα τη Έρευνα και της καινοτομίας. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ανακοίνωση το Σεπτέμβριο του 2012, με την οποία θέτει το πλαίσιο για την συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Η στρατηγική αυτή στην ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάστηκε και από την Επίτροπο Κουίν στην κοινοβουλευτική διάσταση. Υπάρχει ένα τεχνικό θέμα. Διακόπτουμε προσωπικά. Μιλούσα λοιπόν για την στρατηγική μας όσον αφορά τη συνεργασία που παρουσιάστηκε από τον Ρόπερτ Γιάνν Σμιτ στην παρουσίαση που έγινε εδώ στην Επιτροπή σας πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό που θέλω εγώ να σας πω είναι ότι η σύνδεση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Όπως ξέρετε, η σύνδεση με τα διάφορα προγράμματα, με το ίστο για παράδειγμα, είναι πολιτική έκφραση της επιθυμίας να διευρύνουμε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Για πρώτη φορά όμως με τον ορίζοντα 2020 η σύνδεση αναφέρεται στον κανονισμό στο άρθρο 7 του κανονισμού Horizon 2020. Τα ωφέλη είναι πολιτικά, οικονομικά και επιστημονικά. Για τις χώρες ΕΖΕΣ, η σύνδεση με τα ερευνητικά μας προγράμματα διευκολύνει την συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες και προσφέροντας μια νέα αγορά για την έρευνα και την καινοτομία προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των συνδεδεμένων χωρών. οι δύο πλευρές έχουν πρόσβαση και αποφελούνται από την συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο. Για τις προσένταξη χώρες η σύνδεση προσφέρει ένα μηχανισμό με τον οποίο βοηθούν οι χώρες αυτές για να ευθυγραμμιστούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και προετοιμάζεται η πορεία τους προκειμένου να ταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις γείτονες χώρες τα ωφέλη της συνεργασίας συνδυάζονται και με την σημασία που έχει η επιστήμη στην διπλωματία. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω εδώ ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τη σύνδεση σε μια πολιτική ωφέλους μόνο για τους εταίρους μας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφελείται επιστημονικά από τις συμφωνίες αυτές σύνδεσης γιατί προσφέρει στους ερευνητές της Ευρώπης πρόσβαση σε υψηλού επίπεδο επιστημονικές κοινότητες σε άλλες χώρες και βοηθάει την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης επωφελείται και πολιτικά γιατί ενισχύει τις σχέσεις της με τις χώρες που επωφελούνται από την πολιτική αυτή. Επωφελείται επίσης και οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι χώρες οι οποίες είναι γεωγραφικά κοντά στην Ευρώπη είναι και εκείνες οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη σχέση με τις οικονομίες μας. Συνεπώς, ποιοι είναι οι μηχανισμοί της σύνδεσης αυτής. Όπως είπα, ο Horizon 2020 αναφέρεται ρητά στην σύνδεση αυτή. Προηγούμενα προγράμματα ήταν καταρχήν ανοιχτά σε αιτήσει από διάφορες χώρες του κόσμου. Το άρθρο όμως 7 αυτή τη φορά του κανονισμού για τον ορίζοντα 2020 περιορίζει τη σύνδεση σε χώρες της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής. Ιδιαίτερα χώρες ΕΖΕΣ, χώρες διεύρυνσης, γείτονες χώρες και στις χώρες οι οποίες ήδη ήταν συνδεδεμένες στα πλαίσια του ευδέωμου προγράμματος πλαισίου έρευνας. Επιπλέον, από τις γείτονες χώρες, το άρθρο 7, σύμφωνα με την ανακοίνωση για την διεθνή συνεργασία, στην οποία αναφέρθηκα πριν, θέτει κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούν οι χώρες προκειμένου να συνδεδεθούν με το πρόγραμμα αυτό. Τα κριτήρια αυτά είναι καλές ικανότητες επιστημονικές, καλό απολογισμό αν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η συμμετοχή σου σε τέτοια προγράμματα και τρίτον ε, η συμμεταχείριση όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα το καθεστώς σύνδεσης, εμείς προσφέρουμε ενημέρωση στην Επιτροπή σας την Ήτρη, ήδη το Δεκέμβριο το κάναμε και σας έχουμε παρουσιάσει και έναν ενημερωμένο πίνακα τώρα ακριβώς πριν από τη συνεδρίαση αυτή. Αυτό που θέλω να προσθέσω όμως τώρα είναι ότι όλες οι χώρες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το, πρόγραμμα, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο εξέφρασαν την επιθυμία να συνδεθούν και με το πρόγραμμα Horizon 2020. Το θέμα που τίθεται είναι για το Liechtenstein, το οποίο ρητά επί της αρχής ενδιαφέρεται, αλλά το Κοινοβούλιο καταψήφισε την σύνδεση και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον. Για τις υπόλοιπες χώρες ΖΑ ε, και ε, Νορβηγία και Ισλανδία, η διαδικασία έχει προχωρήσει πολύ. Η σύνδεση συμπεριλαμβάνεται σε μια τροποποίηση του πρωτοκόλου 13 όσον αφορά την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την τροποποίηση αυτή πρόσφατα και τώρα περιμένουμε το Συμβούλιο και τις χώρες ΕΖΕΣ τις ίδιες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Προβλέπουμε η σύνδεση να αρχίσει να ισχύει τον Μάιο που μας έρχεται. Όσον αφορά τη σύνδεση τώρα των ε, χώρων προς ένταξη, βασίζεται στις, διαδικασίες, στις συμφωνίες πλαίσιο μάλλον για τη συμμετοχή των χωρών αυτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η προσένταξη χώρες κατά το παρελθόν είχαν συμμετάσχει στο εβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και σύμφωνα με την ανάγκη να αναπτύξουν περισσότερο τις ερευνητικές του δραστηριότητες θα συνεχιστεί και στα πλαίσια του Horizon 2020 η διαδικασία. Πού βρισκόμαστε? Οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί με την ΤΕΟ Ιουσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και την Σερβία. Με την Αλβανία και την Βοσνία Ριζεχοβίνη συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και θα ολοκληρωθούν σύντομα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τελικά η σύνθεση αυτή θα γίνει πλήρης στο τελευταίο τρίμηνο του 2014. Η σύνθεση χωρών τώρα που βρίσκονται γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Όπως λέει και η επιστολή που έστειλε στην κυρία Σαρτόρη, γενικός μας διευθυντή, την 1η Αυγούστου του 2013, οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ξεκίνησαν τον Αύγουστο που μας πέρασε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο έγκαιρα στις 16 Δεκεμβρίου 2013 για το ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας με το Ισραήλ και μετά από την ενημέρωση αυτή το κείμενο της συμφωνίας ε, μονογράφηκε. Περιμένουμε τώρα την τελική απόφαση για τις διαδικασίες και περιμένουμε να υπογραφεί τον Απρίλιο η συμφωνία. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει και με την Μολδαβία. Μάλιστα, ο Γενικό Διευθυντή σήμερα είναι στη Μολδαβία. Η Μολδαβία συνδέθηκε με το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Οπότε βάσει του άρθρου 7 του Horizon 2020 μπορεί, έχει το δικαίωμα να συνδεθεί και με το πρόγραμμα αυτό Horizon 2020. Η Αρμενία επίσης ζήτησε σύνδεση και θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και με την Αλβανία σύντομα για να συζητήσουμε τις προϋποθέσεις για μια πιθανή σύνδεση. Η Ουκρανία επίσης πέρυσι ήδη εξέφρασε την επιθυμία για ενίσχυση του διαλόγου στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να υπάρξει σύνδεση στο μέλλον λοιπόν με την Ουκρανία βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εξαρτάται από τις εξελίξεις στη χώρα αυτή. Έχουμε διάλογο πάντως στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και σχεδιάζουμε να αρχίσουμε συζητήσεις αφού μονογραφεί η συμφωνία να δούμε πώς μπορούν να συνδεθούν καλύτερα με το πρόγραμμα Horizon 2020 και να δούμε αν τελικά μπορούν να συνδεθούν πλήρως ή όχι. Δεν προβλέπουμε όμως συμφωνίες σύνδεσης φέτος με την Ουκρανία. Υπάρχουν τώρα και δύο χώρες όπου εδώ πέρα πρόκειται και αυτόνομες διεθνείς συμφωνίες. Έχουμε, κάνουμε εδώ με την Ελβετία και τις νήσους Φερόες. Ελβετία τα ξέρετε, γιατί όλοι ξέρετε και ο πίτροπος Άντορ έκανε δήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου, στην Ολομέλεια δηλαδή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με λόγια, οι διαπραγματεύσεις ήταν περίπου πλήρης όταν έγινε το δημοψήφισμα για την μετανάστευση στην Ελβετία. Οπότε σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις. Και έχουν για τα νησιά Φαρόε έχουμε ακόμα, είμαστε σε αναμονή να διαπραγματευτούμε την συμμετοχή τους στον ορίζον 2020. Περιμένουμε θα προχωρήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχουν κάποια πολιτικά θέματα που έχουν να κάνουν με μια διεθνής ε, διαμάχη για την αλία που μπορεί να έχουν κάποια επίπτωση όχι για την ίδια την συμφωνία αυτή να συμμετάσχουν στο ορίζον 2020 αλλά για τη χρονική στιγμή εφαρμογή της συμφωνίας που μπορεί να μην εφαρμοστεί αναδρομικά όπως οι άλλες. Θα υποβληθεί πάντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η συμφωνία για έγκριση. Για να κλείσω λοιπόν, περιμένουμε ότι για τις περισσότερες χώρες οι οποίες ζήτησαν να συμμετάσχουν στο ορίζον 2020 η διαδικασία θα τελειώσει πολύ σύντομα ώστε τα περισσότερα από αυτά τα κράτη θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην πρώτη ε, συμφωνία για χορηγήσεις μέσα στο ορίζον 2020. Όπως είπα, προβλέπεται για όλες σχεδόν από αυτές τις χώρες να εφαρμοστούν οι συμφωνίες αναδρομικά από την αρχή του ορίσον 2020, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2014. Και πρώτο Πρωτού κλείσω κάποια λόγια για τις επιστημονικές και τεχνολογικές συμφωνίες. Υπάρχουν 20 τέτοιε συμφωνίες, οι οποίες θα πρέπει να ανανεωθούν όπως είναι σε τακτά διαστήματα, δηλαδή κάθε πέντε χρόνια, αντίθετα με τις συμφωνίες για τη συμμετοχή. Δεν συνδέεται η χρονική στιγμή ανανέωσή τους με το πρόγραμμα πλαίσιο. Να σας αναφέρω λοιπόν ποια είναι η κατάσταση των ανανεωμένων ή ανανεωθησών συμφωνιών. Πρώτα απ' όλα έχουμε ανανεώσει αυτή τη συμφωνία με τη Ρωσία το Φεβρουάριο και το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε αυτό το θέμα με ταχύ τρόπο και σας ευχαριστώ. Επίσης το Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για, την, ε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Μαρτίου και το θέμα πάλι βρίσκεται στο Συμβούλιο. Και μετά υπήρξε η συμφωνία με την Ουκρανία η οποία και αυτή θα ανανεωθεί αργότερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν προς το παρόν για την ε, σύνδεση με το ορίζον 2020 και την ανανέωση τεχνολογικών και επιστημονικών συμφωνιών. Χαίρομαι λοιπόν που είχαμε πάντα πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπω στη συνέχιση του, συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν τώρα αιτήσει να λάβετε το λόγο, ένα λεπτό παρακαλώ καθένας. Ναι, ναι, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλα αυτά που είπατε. Ένα μοναδικό ερώτημα έχω να κάνω. Μάλλον δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι με ποιο τρόπο περιμένω να βάλει τα ακουστικά της η ομιλήτρια με ποιο τρόπο θα δοθούν οι πληροφορίες αυτές σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν προγράμματα τους χρήστες ουσιαστικά, αυτοί που θέλουν να έχουν μια πρόταση. Πότε θα ενημερωθούν από ποιες χώρες μπορούν να υποβάλουν τέτοια προγράμματα. Και το δεύτερο ερώτημα. Στην περίπτωση της Ισλανδίας ή της Νορβηγίας, δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχουν ε, προβλήματα πολιτικά, μπορούν να θεωρηθούν πλήρης εταίροι μας Και το ερώτημά μου τότε το εξή. Για τα σχέδια αυτά όπου συμμετέχουν ε, εταίροι οι οποίοι έχουν ήδη τύχει αναγνώριση στο παρελθόν, οι Κομισιόν και οι λύπτες αποφάσεων θα λάβουν υπόψη και από ποιες χώρες έρχονται αυτοί οι οποίοι υποβάλλουν σχέδια και προγράμματα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ε, προτιμούμενες ή μη προτιμούμενες ή έχουν όλες το ίδιο δικαίωμα. Η κυρία Κωστέτ. Πάρα πολύ σύντομα, λέει η κυρία κυρια παρα πολυ συντομα Υπάρχει μια συμφωνία με το Ισραήλ. Θα ήθελα να ξέρω όταν υπάρχουν ερευνητικά σχέδια τα οποία έχουν σαν έδρα τους χώρους των ε, κατεχωμένων από το Ισραήλ ε, εδαφών αν μπορούν να επιδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάτε και για την Ελβετία που είναι δύο ρηξιές από το σπίτι μου. Οι Ελβετοί επιστήμονες έχουν πάρει πάρα πολύ σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007. Τώρα ξέρουμε ότι όλα αυτά έχουν ανασταλεί, αλλά μήπως έχετε κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις να μου δώσετε για το θέμα αυτό. Περιμένω ότι οι Ελβετοί ερευνητές θα βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι θέλει κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Επομένως, σας ξαναδίνω το λόγο για να απαντήσετε. Στην Διευθύντρια Ρούσο έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με την ενημέρωση έχουμε ένα δίκτυο που λειτουργεί σωστά Έχουμε τα εθνικά σημεία επαφής σε όλα τα κράτη-μέλη και στις συνδεδεμένες χώρες στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 και χρησιμοποιούμε τα δίκτυα αυτά συνεργαζόμενοι και με τις αρμόδιες επιτροπές και στα πλαίσια των προγραμμάτων τα οποία είναι σε λειτουργία σήμερα. Έχουμε επίσης ε, ε, τη νέα ηλεκτρονική θύρα ενημέρωσης. Υπάρχουν επίσης τα κράτη-μέλη και στις συνδεδεμένες χώρες ε, κάποιες ημερίδες για την εκκίνηση του προγράμματος Horizon 2020. Είναι σημαντική η ενημέρωση και κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Φυσικά αυτό είναι και προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Ευρώπη 2020 και η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του καθενός από με μεμονωμένα είναι σημαντική. Για την Ισλανδία και την Νορβηγία και τα ισότιμα δικαιώματα συμμετοχής είπα ήδη ότι όταν υπάρχουν τρίτες χώρες οι οποίες συνδέονται με το Horizon 2020 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα κράτη-μέλη, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα κράτη-μέλη και ανήκουν στον σκληρό πυρήνα θα έλεγα των ε, χωρών που αποτελούν ε, τα διάφορα κονσόρτια. Το ότι είναι συνδεδεμένες χώρες όμως δεν τους δίδουν κυρίαρχη θέση επί των άλλων απλά έχουν τα ίδια δικαιώματα. σαν τα κράτη-μέλη και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσω και στην κυρία Γκροστέτ σχετικά με την Ελβετία. Η Ελβετία τώρα δεν μπορεί στην παρούσα φάση να συνδεθεί με το Horizon 2020 αλλά μπορεί να συμμετέχει στο σύνολο του προγράμματος αυτού σαν τρίτη χώρα γιατί το Horizon 2020 είναι ανοιχτό στη συμμετοχή των τρίτων χωρών και η Ελβετία επειδή δεν είναι πλέον συνδεδεμένη, δεν θεωρείται έτσι, συμμετέχει στο πρόγραμμα όχι όπως τα κράτη-μέλη αλλά ως τρίτη χώρα. Αυτή ήταν η κατάσταση έτσι και αλλιώ και στο πέμπτο ε, πλαίσιο έρευνας πριν από τη Συμφωνία Σύνδεσης. Είναι σημαντικός εταίρος η Ελβετία, το υπογραμμίσατε και το υπογραμμίζω και εγώ. <clears throat> Να πω ότι οι ελβετικές αρχές που ασχολούνται μετά της έρευνας ανησυχούν και ψάχνουν να βρουν δυνατότητες χρηματοδότησης για να μπορέσουν να βοηθήσουν στη συμμετοχή των ερευνητών στο Horizon 2020. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι στην παρούσα φάση οι διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί, αλλά οι συζητήσεις με τους Ελβετούς συνεχίζονται και μάλιστα αύριο ο δεύτερος Γενικός Διευθυντής μας, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, θα συναντηθεί με τον αρμόδιο γραμματέα για την έρευνα. Για τα κατεχόμενα τώρα, και με τη συμφωνία με το Ισραήλ εμείς εφαρμόσαμε τους προσανατολισμούς τις οποίες η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δημοσίευσε τον προηγούμενο Ιούνιο για την αντιμετώπιση των οντοτήτων όχι μόνο έρευνας που υπάρχουν στα κατεχόμενα. Οι οντότητες αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Horizon 2020 ε, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ελπίζω να απάντησα. Καλό, σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν το τμήμα αυτό της συνεδρίασης. Το ανοιχτό, το δημόσιο κομμάτι της συνεδρίασής μας. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και την κυρία Ρούσο για την παρουσία της και για τα στοιχεία που μας έδωσε, χρήσιμη. Εμείς δεν θα έχουμε δυνατότητες να συναντηθούμε εκ νέου μαζί σας, αλλά μετά από τις νέες εκλογές θα υπάρξει, ελπίζω, καλή συνεργασία με σας. Σας ευχαριστώ κυρία Ρούσο λοιπόν και στο επανειδήν. Α, υπενθυμίζω επίσης στους συναδέλφους πριν φύγουν ότι σήμερα το απόγευμα σε αυτή την αίθουσα το απόγευμα θα γίνει μια άλλη συνεδρίαση και γι' αυτό σας παρακαλώ να μην αφήσετε τα έγγραφά σας στην αίθουσα. Αν και έχουμε αύριο την συνεδρίασή μας την τακτική εδώ. Γι' αυτό σας παρακαλώ να πάρετε μαζί σας όλα τα έγγραφα τα οποία σας αναλογούν. Αύριο το πρωί λοιπόν γνωρίζετε ότι στις 9 θα ξεκινήσουμε 9 με 10 με μια συνεδρίαση εδώ σε αυτή την αίθουσα και από τις 10 και μετά θα ψηφίσουμε και πριν ψηφίσουμε θα φωτογραφηθούμε. Σας ευχαριστώ όλους στο επανειδήν παρακαλώ να παραμείνουν μόνο οι συντονιστές.